Okay, dear colleagues, to uh, Συνάδελφοι, καθίστε. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Εσεί, οι δύο που μιλάτε, Σα παρακαλώ να σταματήσετε. Μετά θα έχουμε χρόνο για κουβέντα. Με μεγάλη μα χαρά, λοιπόν, σας καλωσορίζουμε, κύριε Υπουργέ, Υπουργό Υγεία τη Κροατία είναι εδώ μαζί μα ε, και εκ μέρου τη Κροατική Προεδρία. Φυσικά, γι' αυτό λοιπόν θα σα δώσουμε περίπου 10. 12 λεπτά έτσι ώστε να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες ε, της Κροατίας για τον τομέα της υγεία, το επόμενο εξάμεινο και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου, ελπίζω λοιπόν να φορέσετε τα ακουστικά σας. Για τα επόμενα 10 λεπτά λοιπόν θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Κροατίας, ενός ε, νέου κράτους μέλους που ε, έχει αναλάβει την πρώτη του Προεδρία. Στην Κροατία, λοιπόν, έχουμε δώσει έμφαση σε δύο τομείς. Ο πρώτος αφορά την δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων. Στην Κροατία έχουμε μεγάλη εμπειρία την οποία θέλουμε να μοιραστούμε. Εμπειρία ιδιαίτερα στην δωρεά οργάνων. Και επίσης θα θέλαμε να μοιραστούμε την εμπειρία μας ε, πάνω στην μεταμόσχευση οργάνων που είναι κάτι που σώζει ζωές όπως ξέρετε. Σήμερα επίσης θα σας μιλήσω για κάτι που αφορά άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και ενώ τη γύρανση του πληθυσμού. Πάνω από το 25% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άνω των 65 ετών. Και όπως γνωρίζετε, όσο μεγαλώνει κανείς, αυξάνονται και οι περιπτώσεις ε, να, να νοσήσει κάποιος ε, από διάφορες ασθένειες, ε, καρκίνους κτλ. Τούτο φυσικά συνεπάγεται αυξήσεις δαπανών για τον τομέα της υγείας. Θα ήθελα λοιπόν με την άδειά σα να αναφερθώ πρώτα στη μεταμόσχευση οργάνων. Πριν από αρκετά χρόνια στην Κροατία ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε εντατικά και να τρέχουμε διάφορα προγράμματα δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων. Έχουμε εμπειρία 40 ή 50 ετών, τότε που ξεκινήσαμε δηλαδή και τα προγράμματα αυτά. Έχουν σωθεί πάρα πολλές ζωές, διότι στο παρελθόν οι άνθρωποι πέθαναν επειδή δεν υπήρχαν αρκετά όργανα για μεταμόσχευση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για το θέμα αυτό ενημερώνοντάς τους ότι μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους εκ των προτέρων έτσι ώστε να γίνουν δωρητές οργάνων και να μπορέσουν λοιπόν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Σε περίπτωση που αποβιώσουν και τα όργανα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αν δούμε τώρα το μέσο όρο δωρητών οργάνων στην Κροατία, θα παρατηρήσετε ότι οι δωρές οργάνων έχουν διπλασιαστεί και είναι κατά πολύ ψηλότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεταμόσχευση οργάνων, στην Κροατία έχουμε παρατηρήσει πολλά ωφέλη για τους ασθενείς. Και τον Απρίλιο θα έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες μας και να διοργανώσουμε άλλη μια καμπάνια ευαισθητοποίησης ε, των πολιτών. Οι γιατροί μας επίσης θα είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Και θα θέλαμε λοιπόν να παροτρύνουμε και τους ε, γειτονές μας έτσι ώστε να μας ακολουθήσουν σε αυτή την πρωτοπορία. Υπάρχουν ορισμένα όργανα που μπορούν να αντικατασταθούν από τεχνητά μέρη. Όμως όχι όλα. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξε ένα πρόγραμμα μεταμόσχευσης οργάνων ζώων σε ανθρώπους και ο ίδιος προσωπικά εργάστηκα πάνω σε αυτό το πρόγραμμα υπό τον καθηγητή David Cooper όπου μελετήσαμε τις ε, αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος σε αυτές τις μεταμοσχεύσεις ε, οργάνων. Θεωρούμε λοιπόν ότι εάν προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε τους πολίτες να γίνουν δωρητές οργάνων υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλο αυτό θα γίνει με τρόπο ηθικό και ε, συμβατό με τη διοντολογία, τότε είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να σωθούν ζωές μέσω της μεταμόσχευσης. Γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, ε, να γίνει ένας διάλογος με στόχο να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας σκοπεύουμε επίσης να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Θα διοργανώσουμε λοιπόν μία ε, ημερίδα στο Ζάγκρεμπ, ένα συνέδριο για ε, το κόστος μιας ασθένειας. Ορισμένες ε, ασθένειες έχουν πολύ ψηλό κόστος για τον τομέα της υγείας. Επίσης, ε, θα μιλήσουμε και για τα προγράμματα διάγνωσης, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Και εδώ χρειάζεται διάλογος, ανταλλαγή εμπειρίας, διότι έχουμε παρατηρήσει πως ε, υπήρξαν προγράμματα τα οποία δεν πήγαν καλά ακριβώς ε, διότι δεν ε, υπήρξε έντονη αντίδραση. Για παράδειγμα, προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης ε, διαφόρων μορφών καρκίνου του τραχύλου, ας πούμε. Είχαν γίνει κάποια προγράμματα πρόληψης και ελέγχου που έτρεξαν περίπου για 13-14 χρόνια, όμως δεν είχαν μεγάλη απήχηση και δεν ήταν επιτυχή. Στην εθνική μας στρατηγική λοιπόν για την ε, έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση του καρκίνου δώσαμε έμφαση στον έλεγχο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να συνεργαστούμε και με τα άλλα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αυξηθούν αυτά τα προγράμματα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος ε, Υγείας έχει μάλιστα συμπεριλάβει στη στρατηγική του προγράμματα έγκαιρης ε, διάγνωσης καρκίνου. Είναι μια τεράστια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες, να συζητηθεί το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, έτσι ώστε να μειωθούν τα κρούσματα καρκίνου. Είναι πολύ σημαντικό ε, τέτοιες ασθένειες να εντοπίζονται όσο το δυνατόν συντομότερο έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να, έχουν, να υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Όσο πιο αρχικό είναι το στάδιο λοιπόν ε, που εντοπίζουμε μια ασθένεια, τόσο πιο καλή πρόγνωση. Υπάρχουν κάποια προγράμματα ελέγχου διαγνωστικού για ορισμένες μορφές καρκίνου. Για παράδειγμα, ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου και είναι περίπου στην τρίτη, τέταρτη ε, θέση σε ό,τι αφορά τους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το 15% των ε, ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμα να επιβιώνουν. Όμως, ε, αν εντοπιστεί νωρίς, μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία και να σώσει χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει στην Κροατία να χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα που στόχο έχει καπνιστές μεταξύ 50 και 70 ετών ή άτομα τα οποία έχουν στην οικογένειά τους ιστορικό καρκίνο του πνεύμονα. Καλούμε λοιπόν τα άτομα αυτά για διαγνωστικό έλεγχο έτσι ώστε να εντοπιστεί αυτός ο καρκίνος το συντομότερο δυνατό και να μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Θα σας ενημερώσουμε λοιπόν στο συνέδριο στο Ζάγκρεπ για τα ευρήματά μας ε, σχετικά με αυτό και φυσικά θα σας ενημερώνουμε ανατρίμηνο για τις εξελίξεις. Αν η εμπειρία μας ε, είναι θετική, ελπίζουμε εσείς να λάβετε υπόψη τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει στον τομέα αυτό και να λειτουργήσουμε υποδειγματικά για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια μεγάλη ηλικία και να ζούμε καλά θα πρέπει να αλλάξουν αρκετά. Θα πρέπει ο τρόπος ζωής μας να είναι υγιής και εδώ έρχομαι να αναφερθώ στα διάφορα προγράμματα ηλεκτρονικής υγείας, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω ευχαριστώντας σας για την προσοχή. Είμαι στη διάθεσή σας για ε, οποιαδήποτε ερώτηση και φυσικά για οτιδήποτε ξέχασα να πω. Σας ευχαριστώ. Thank you very much for having... Σας ευχαριστώ. Εκθέσατε τις προτεραιότητά σας με ξεκάθαρο τρόπο. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πιτελίζα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα τώρα να πάρω την ευκαιρία για να καλωσορίσω μία ομάδα νέων από τη χώρα μου, καλεσμένη ενός άλλου συναδέλφου, νέοι οι οποίοι ασχολούνται με την ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Τώρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Φυσικά η δωρεά οργάνων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα. Πρέπει να το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς. Πριν από μερικά χρόνια βελτιώσαμε την νομοθεσία σχετικά με την ε, δωρεά οργάνων. Η νομοθεσία αυτή επέτρεψε να γίνεται διανομή οργάνων από κράτος μέλος σε κράτος μέλος έτσι ώστε να μην πηγαίνει καμία ευκαιρία χαμένη και να μπορούν να υποφεληθούν όλοι οι πολίτες από τη δωρεά οργάνων. Θα ήθελα λοιπόν να διευρυνθούν αυτές οι προσπάθειες και αυτές οι συμφωνίες ανταλλαγής. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει μια αντίστοιχη συμφωνία με την Αυστρία για ανταλλαγή οργάνων. Όμως ε, αυτές οι διμερείς συμφωνίες δεν ισχύουν ε, για όλα τα κράτη. Για παράδειγμα, με την Πολωνία δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Για την ομάδα μου επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην συνολική προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στις μονομένες προσπάθειες των κρατών μελών. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα του παιδικού καρκίνου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ε, οδυνηρό τόσο για το παιδί όσο και για την οικογένεια. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν προσπάθειες ε, για να υπάρχουν φάρμακα για τον καρκίνο, για όλους. Έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το, πρόβλημα αυτό ε, πιο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι ζούμε την εποχή της πληροφορίας. Αλλά δυστυχώς η παραπληροφόρηση και τα fake news τα λεγόμενα στον τομέα της υγείας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει έτσι ώστε να προωθήσουμε ε, ε κάποιες ιδέες για καλύτερη και πιο υγιεινή ζωή η σωστή ετικετοθεσία, η σωστή ενημέρωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή κάνει προσπάθειες για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ξέρουμε ότι το 40% των καρκίνων θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί είναι σαφές ότι ε, θα πρέπει να ληφθούν το ταχύτατο μέτρα. Επίσης έχουμε και το θέμα της αντίστασης στα μικροβιωτικά, στα αντιβιωτικά. 25 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από μία μη αποτελεσματική χρήση των αντιβιωτικών ουσιών. Υπάρχουν πολλοί τομείς ε, στους οποίους μπορεί να ληφθούν μέτρα. Είναι μια διατομεακή πολιτική και δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στο θέμα της υγείας. Θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη προσπάθεια από πλευράς μας και στον τομέα της ασφάλειας και στον τομέα της κατοικίας και στον τομέα της διατροφής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Υπουργό. Σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίσατε ε, την υποφασιστικότητά σας για την καταπολέμηση του καρκίνου και την επιθυμία που έχετε να κινητοποιηθούμε στον τομέα της πρόληψης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την προηγούμενη εβδομάδα το λεγόμενο Green Deal. Περιλαμβάνονται πάρα πολλά μέτρα πρόληψη στον τομέα της υγείας. Ένα από τα μέτρα σχετικό με τη διατροφή είναι η βελτίωση των τροφίμων, των προϊόντων τροφίμων μέσω της συσκευασίας και της ε, ετικετοθεσίας. Το λεγόμενο Nutri-Score είναι θα έλεγα μια ιατρική απόδειξη η οποία δείχνει ότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα μειωθεί η θνησιμότητα για τις χρόνιες παθολογίες κατά 3%. Είναι κάτι το οποίο είναι κατανοητό, ιδιαίτερα για τους λιγότερο ευνοημένους οικονομικά και κοινωνικά πληθυσμούς. Είναι ένα μέσο το οποίο θα βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της υγείας και είναι και μια ανάγκη την οποία έχουν οι καταναλωτές. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις οι οποίες έχουν ε, μάλιστα οδηγήσει και σε ένα ψήφισμα με 90.000 υπογραφές έτσι ώστε το Nutri-Score να καταστεί υποχρεωτικό για όλα τα ευρωπαϊκά τρόφιμα. Να μου πείτε λοιπόν κύριε Υπουργέ ποια είναι η άποψή σας για την στρατηγική Farm to Fork από το αγρόκτημα στο Πυρούνι ε, και να μας μιλήσετε επίσης και για το θέμα αυτό του Nutri-Score που θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τους πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Παουλούς. Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε, τη σημασία δηλαδή ε, του να κάνουμε βήματα επιτέλους για την καταπολέμηση του καρκίνου. Και χαίρομαι που και η συνάδελφος από τους σοσιαλιστές αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και όχι μόνο της θεραπείας. Η πρόληψη είναι φθηνότερη από την θεραπεία και ε, πράγματι αποφεύγονται τρομακτικές πιέσεις στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ε, ποιος είναι ο ρόλος σας για ένα μη τοξικό περιβάλλον. Το μη τοξικό περιβάλλον είναι τμήμα του 7ου προγράμματος πλαισίου, δεν έχει ακόμα προωθηθεί θεωρείται περιβαλλοντικό απλά θέμα, ενώ δεν είναι μόνο, είναι θέμα υγείας πριν απ' όλα. Ένα παράδειγμα είναι οι ενδοκρινοκοί ε, διαταρακτές. Είναι ορμόνες που επηρεάζουν ε, ε, τις αντίστοιχες ορμόνες στο ανθρώπινο σώμα και δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία των οργάνων, μπορεί να οδηγήσουν και σε καρκίνους, ακόμα και σε πολύ μικρές ποσότητες. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, μια συγκεκριμένη στρατηγική για τους ενδοδιακρινικούς ε, ε, διαφταράκτες, Συνεπώς λοιπόν αντιμετωπίζεται ένα προϊόν που περιέχει ας πούμε ε, τέτοιες ουσίες με διαφορετικό τρόπο από ότι ένα ζυζανιοκτόνο που μπορεί να περιέχει τέτοιες ουσίες. ένα τέτοιος ε, διαταράκτης είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να περιλαμβάνεται σε υλικά στα οποία ε, είμαστε σε συνεχή σωματική επαφή, το πάτωμα, ε, τα παιδιά μπορεί να τρώνε στο πάτωμα. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν σκοπεύετε να κάνετε κάτι στον τομέα αυτό έτσι ώστε να υπάρξει μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μη τοξικό περιβάλλον. Ε, πήρατε το χρόνο δύο μελών ε, για τους πρασίνους. Από τα ID δεν έχουμε μιλητή. Με το ECR, κυρία Κονσίνσκα, αλλά δεν είναι εδώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερως που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά θέματα εδώ μαζί σήμερα. Εγώ θα ήθελα να σας θέσω δύο πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Μάλλον ελήψη χρόνου. Δεν μας είπατε τι προτίθεστε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε τη γύρανση του πληθυσμού. Ποια δέσμη μέτρων θα μπορούσατε να προτείνετε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Και ποιες είναι οι απειλές που έχουμε εδώ. Η Προεδρία σας τι θα κάνει για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Θα περιμένουμε κάποια πρόταση. Τι προσέγγιση θα έχετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδατε ότι περισσότεροι ομιλητέ ρώτησαν για τον καρκίνο και πώ θα τον καταπολεμήσουμε. Στην Επιτροπή μα ψηφίσαμε μια σύσταση για την αύξηση των κονδυλίων για την ε, καταπολέμηση του καρκίνου. Κάναμε και ακρόαση με, με τον Επίτροπο Υγείας, αλλά δεν πήραμε συγκεκριμένες ε, απαντήσεις για το πώς ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να καταπολεμήσει τον καρκίνο. Όλα αυτά συνδέονται και με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάποιες ιδέες και προτάσεις. Ευχαριστώ. Γκουε. Για να κλείσουμε τον πρώτο γύρο. Παρακαλώ. Η κυρία Μόντι. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στην Κροατία για την πρώτη της Προεδρία. Εγώ είμαι Φιλανδή. Η Φιλανδία είχε την προηγούμενη την Προεδρία το προηγούμενο εξάμεινο. Ξέρω λοιπόν ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καλή επιτυχία λοιπόν σας εύχομαι. Η Κροατία πώς θα αντιμετωπίσει τις ασθένειες που προκύπτουν από ε, την κακή ποιότητα του αέρα, της ατμόσφαιρας. Πώς θα αντιμετωπίσετε την ε, χρήση ε, ρηπαντών της ατμόσφαιρας και ζανιοκτώνων που χρησιμοποιούνται ευρέω ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα με άλλου συναδέλφου, ήθελα και εγώ να ρωτήσω για του ενδοκρινικού ε, διαταράκτε, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο καθότι πλήττουν ε, ε, την ανθρώπινη υγεία με πολλούς και διάφορους τρόπους. Η επισήμανση των τροφίμων, πώς θα προωθήσουμε τις καλές πρακτικές σε αυτό το τομέα και πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα δεν θα συμπεριλαμβάνουν ε, ε, υλικά που πλήττουν την ανθρώπινη υγεία. Μίλησε για τα προληπτικά μέτρα, πολύ θετικά. Όλα αυτά που αναφέρατε επηρεάζουν την υγεία. Μετά, πώς ε, βλέπετε την προώθηση μιας χορτοφαγικής δίαιτας ή ακόμα και vegan διατροφής γιατί βλέπουμε ότι ο, ο κλάδος ε, της βιομηχανικής παραγωγής κρέατος ε, κάνει το παν για να αποτρέψει τον κόσμο από το να στραφεί σε μια τέτοια διατροφή που θα βασίζεται στα φυτά. Πώς θα προωθήσετε εσείς όμως αυτή την ε, πρακτική που είναι σημαντική. Έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε στο πρώτο γύρο. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ για όλα σας τα ερωτήματα. Από τις ερωτήσεις σας συμπεραίνω ότι έχουμε την ίδια προσέγγιση και τις ίδιες ανησυχίες. Και μου φαίνεται ότι έχουμε και το ίδιο όραμα, την ίδια προσέγγιση ό,τι αφορά την επίλυση του προβλήματος. Δεν γίνεται να στρέψουμε το βλέμμα μακριά από την πραγματικότητα. έχουμε παράγοντες που μπορούν να ζημιώσουν την ανθρώπινη υγεία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνήσουμε γιατί ένα εκατομμύριο ζωές χάνονται κάθε χρόνο από τέτοιου είδους ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της ε, κρατικής προεδρίας θα εξετάσουμε και θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα φυσικά και δεν θα τα επιλύσουμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προαγάγουμε τον διάλογο. Δεν θα αγνοήσουμε κανένα ζήτημα. Θα συζητήσουμε τα πάντα με επιστημονικό τρόπο και δεν θα ασκούμε πιέσεις σε κανέναν, ανεξάρτητα από το τι θέλει η μία ή η άλλη βιομηχανία. Όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας ε, στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τις ε, μεταμοσχεύσεις, υπόθηκε ότι κάποιες χώρες ε, συνεργάζονται θετικά με τη Γερμανία για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, ενώ σε άλλες δεν επιτρέπεται. Αυτή, αυτό το δίκτυο των ευρωμεταμοσχεύσεων, αν θέλετε, θα μπορούσε να επεκταθεί, ούτως ώστε όλα τα κρατημέλη να συμμετάσχουν στο δίκτυο. Γιατί έτσι πραγματικά μπορούν να σωθούν χιλιάδες ε, ζωές κάθε χρόνο. Και εγώ μιλώ από επιστημονικής, από πολιτικής, ιατρικής άποψης. Αιτιολογείται το να συμμετάσχει κανεί σε αυτό το δίκτυο, να ε, προαγάγει έτσι τις ε, μεταμοσχεύσεις. Για τον καρκίνο. Είπα και πριν ότι πρόκειται για μια τεράστια παγκόσμια πρόκληση. Το μέλλον έγκυται στην ανοσοθεραπεία και στην ε, γενετική θεραπεία, γονιδιακή μάλλον. Γιατί εκεί θα υπάρχουν σίγουρα ωφέλη που θα προκύψουν από τέτοιες θεραπείες. Μόνο αν εργαστούμε από κοινού λοιπόν, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα προχωράμε από κοινού και δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις. Εμείς λοιπόν προωθούμε αυτό το ζήτημα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μαζί πρέπει να μιλήσουμε στον κλάδο και να ε, καταφέρουμε όσο δυνατόν χαμηλότερε τιμέ για τι θεραπείε του καρκίνου. Και να επισημάνω ταυτόχρονα ότι υπάρχουν τεράστιε αυξήσει ε, τιμών στον τομέα του φαρμάκου. Εκεί υπάρχουν τεράστια κέρδη λοιπόν. Μόνο μαζί μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την τάση. Και μέσα στα επόμενα χρόνια, 10 χρόνια, να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει σημαντική πρόοδος. Γιατί μπορούμε να περιμένουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στην επόμενη δεκαετία. Όπως και να έχει, κάθε φορά που μιλά κανείς για τη θεραπεία, γνωρίζει τις δυσκολίες. Γι' αυτό και πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πρόληψη. Όλα αυτά στα οποία εκτιθέμεθα αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες να νοσήσουμε από διάφορες ε, παθήσεις, χρόνιες και μη. Ο τρόπος ζωής μας λοιπόν επηρεάζει τα πράγματα. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι παράγοντες στο περιβάλλον ή στα τρόφιμα που ενδέχεται να μας μειώσουν, θα πρέπει να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό θα μας επιτρέψει να σώσουμε και πάλι ζωές. Πρέπει να υπάρχει διάλογος, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή λύση, ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο για τέτοιου είδους ενέργειες. Φυσικά κάθε χώρα θα πρέπει να έχει ένα τοξικολογικό ε, κέντρο που θα αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις και θα εντοπίζει τι ακριβώς υπάρχει μέσα στα προϊόντα αν υπάρχει κάποια ουσία που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Όπω και να έχει, πρέπει να υπάρχει σαφή επισήμανση στα τρόφιμα, ούτω ώστε οι καταναλωτέ να γνωρίζουν ακριβώ τι αγοράζουν. Αν αγοράζουν ακόμα και κάτι φθηνό σαν προϊόν, να είναι σίγουροι ότι δεν θα καταναλώσουν κάποια επιζήμια ουσία. Όλους μας προβληματίζει το θέμα του περιβάλλοντος Και εγώ από πλευράς μου κάνω ό,τι μπορώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα συμμετάσχουν όλες οι πλευρές, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, για να έχουμε όσο γίνεται χαμηλότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον από την χρήση φαρμάκων. Ένα από τα πρώτα γρήγορα βήματα που μπορούμε να κάνουμε κάποιες ε, χώρες ήδη το έχουν επιλέξει, έχει να κάνει με την αντιμικροβιακή αντίσταση. Όταν υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση αντιβιωτικών, αυτό ενδυναμώνει ορισμένα στελέχη ιών που και πάλι μπορούν να στοιχήσουν σε ανθρώπινες ζωές. Και πρόκειται για ε, ζωές που χάθηκαν ακόμα και αν οι ασθενεί δεν είχαν κάποια τρομερή νόσο. Απλώς ε, μπήκα στο νοσοκομείο και κόλλησαν ένα, ένα τέτοιο ισχυρό στέλεχος ιού εξαιτία τη αντιμικροβιακή αντίσταση. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση σε αυτό το τομέα. Και μετά την Κροατία, ελπίζω και η Γερμανία να συνεχίσει τις προσπάθειές ε, μας για τη διάρκεια της δικής της Προεδρίας. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην τύχη λοιπόν. Θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να προγραμματίσουμε τις ε, προσπάθειές μας. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που δεν ε, απάντησα. Όταν μιλούμε για τοξίνες στο περιβάλλον και ζενεκτόνα που καταναλώνουμε μέσω της τροφής, <coughs> πρέπει να είμαστε σε θέση να τα εντοπίσουμε. Γιατί πράγματι καταστρέφουν το Ακόμα και το άγχος, ακόμα και χημικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ανθρωπίνη υγεία. Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε χημικά που καταλήγουν ε, στα οστερικά όργανα του ανθρώπου, διαταράσουν απόλυτα την ισορροπία του οργανισμού και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλές ε, και πολύ άσχημες ε, παθήσεις. Και εγώ ως ε, γαστεντρολόγος τα έχω δει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ακόμα και νέους ανθρώπους, 20-30 χρονών, να λαμβάνουν μια τέτοια διάγνωση. Κάτι πραγματικά θλιβερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και το νοσοποιητικό και το ενδοκρινικό επηρεάζονται πάρα πολύ και εδώ οι χημικές ουσίες σίγουρα επηρεάζουν τον οργανισμό ε, μέσω των τροφίμων ή ακόμα και της ακτινοβολίας, που είναι κάτι το οποίο δεν συζητούμε συχνά, ίσως όμως θα έπρεπε. Τώρα, για τη γύρωση του πληθυσμού, τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα υπάρξουν φυσικά γρήγορες λύσεις, αλλά μπορούμε να κάνουμε μία διακήρυξη ε, όλα μαζί τα κράτη-μέλη. Να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις ε, συνήθειες του κόσμου. γενικά να γίνουμε πιο δραστήριοι. Υπάρχουν υψηλότερα επίπεδα παχυσαρκίας και στα παιδιά σήμερα σχέση με το παρελθόν. Πρέπει λοιπόν να τους ε, εκπαιδεύσουμε για το τι πρέπει να τρώνε και τι να αποφεύγουν. Στο δικό μου πεδίο εμείς εξετάζουμε όλα τα συστήματα που ενδέχεται να επηρεαστούν και προσπαθούμε να δούμε ποια μέτρα μπορούμε να υλοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Συμφωνώ λοιπόν ότι σε όλες τις ετικέτες τροφίμων, πέραν της χημικής σύστασης, θα πρέπει ξεκάθαρα να αναφέρεται, και η θερμιδική αξία του προϊόντος. Για να ξέρουμε ως καταναλωτές ακριβώς τι παίρνουμε, τι καταναλώνουμε και τι κινδύνους ενέχει αυτό το προϊόν. Τώρα για την χορτοφαγική διατροφή, σίγουρα πρέπει να το συζητήσουμε στο πλαίσιο μιας ε, ε, υγιεινής διατροφής. Θα μπορούσε λοιπόν να προαχθεί μια τέτοια προσέγγιση ως προς τη διατροφή. Αλλά το να είναι κανείς χορτοφάγος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ε, δεν υπάρχουν ζυζανιοκτώνα ή άλλε βλαβερέ ουσίε στα τρόφιμα που καταναλώνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να διευκρινίσετε κάτι εδώ. Ε, την ερώτηση που τέθηκε από το farm to fork Ε, τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις και για τους διαταράκτες και για τις ε, των προϊόντων, τροφίμων. Ε, ποια θέματα είναι αυτά στα οποία θα αναλάβετε την πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια της δικής σας Προεδρία θα παρουσιάσετε αυτό το πρόγραμμα και είναι κάτι το οποίο ε, αφορά και στους Υπουργούς Υγείας και όχι μόνο τους Υπουργούς Γεωργίας και τους Υπουργούς Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ γιατί με την ερώτηση αυτή πράγματι θυμήσατε τη σημασία που έχει το πρόγραμμα αυτό. Πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι. Η πρωτοβουλία αυτή από το αγρόκτημα στο πυρούνι, στο τραπέζι, είναι κάτι που πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Ε, θα προτείνει η Κροατική Προεδρία μια εγκάρσια στρατηγική έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα όχι μόνο σαν γεωργικό αλλά σαν θέμα υγείας. Δημιουργούνται ασθένειες, θάνατοι και το τίμημα το πληρώνουμε όλοι και γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν στη μεγάλη σημασία που έχει το σχέδιο αυτό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο των κρατών μελών, αυτό θα είναι μια μεγάλη πρόοδο στον τομέα της υγείας περνάμε στον δεύτερο γύρο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ε, θα είμαστε σύμμαχοι εναντίον του καρκίνου τα επόμενα χρόνια. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει το θέμα των τοξικών χημικών δεν είναι μόνο να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά και τον εαυτό μας. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε για την καταπολέμηση του καρκίνου ε, μέσω της καταπολέμησης των χημικών τοξικών. Δεύτερη ερώτηση. Η διάκριση ανάμεσα στις θεραπείες, της παιδιατρικές και στις θεραπείες των ενηλίκων και θα ήθελα εδώ να μου πείτε πώς βλέπετε τις διακρίσεις ανάμεσα στις ηλικιακέ αυτές ομάδες. Και να πω επίσης ότι αυτό το οποίο ελείπει και είναι το τρίτο θέμα είναι η μετά την επέμβαση αντιμετώπιση των προβλημάτων των καρκινοπαθών. Ο Τίμο Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, στον ε, τομέα της ιατρικής ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εδώ. Όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτό, διότι μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό. Επίσης, η HTA η αξιολόγηση της τεχνολογίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να υπάρξει μια προσέγγιση όλων των εθνικών συστημάτων υγείας έτσι ώστε να έχουν όλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και νέες ε, θεραπείες. Έχει γίνει μια σχετική πρόταση πριν από δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από τις 14 ε, Φεβρουαρίου του 2019 το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του σε αυτό το θέμα, έχει όμως κολλήσει στο Συμβούλιο και δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ρωτήσω, η δική σας Προεδρία τι προτίθεται να κάνει έτσι ώστε να βοηθήσει για να ξεκολλήσει το θέμα αυτό από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται έτσι ώστε να επωφεληθούν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης ε, με ευκολότερη πρόσβαση σε φάρμακα. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια συγκεκριμένη λύση για αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε προκαταβολικά γιατί θα είστε η πέμπτη Προεδρία που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα από τότε που ξεκίνησε το διέξοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Renew. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να συνεχίσω και εγώ λέγοντας ότι υπάρχει όντως πρόβλημα στην διαθεσιμότητα των φαρμάκων. Ε, το πρόβλημα αυτό υπάρχει παντού, ακόμα και στις κατοχώρες. Το 2002 μέχρι το 2004 υπήρχε έλλειψη φαρμάκων για αρκετούς μήνες ή ακόμα περισσότερο. Το 2019 οχταπλασιάστηκε ο αριθμός αυτός, δηλαδή 700-800 διαφορετικά ε, φάρμακα ήταν σε έλλειψη. Και αυτό λοιπόν ε, καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μεμονωμένα. Ο Υπουργό Υγεία μα, ε, λοιπόν, ο Μπρούνο Μπράουνς, έχει προτείνει να υπάρχει ένα απόθεμα φαρμάκων αρκετό για πέντε μήνε στι κατοχώρε. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι οι ειδικοί μάλιστα λένε ότι μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα αυτό θα επιδεινωθεί. Οι ειδικοί λοιπόν θεωρούν ότι πρέπει να αποκτήσουμε ξανά τις πηγές τις πρώτες ύλε για την παραγωγή αυτών των ε, φαρμάκων, έτσι ώστε να μπορούμε να ε, κατασκευάζουμε αυτά τα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην εξαρτώμεθα από τρίτες χώρες. Εσείς ε, λοιπόν ε, τι προτίθεστε να κάνετε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει το λόγο ε, κάποιο από τους πράσινους ή από το ID. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του ECR. Ή δεν έχει έρθει. Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Η κυρία ερθει ακομα η κυρια να εκ μέρου τη Γκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ως συνέχεια αυτών που είπαν οι συνάδελφοι λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να πω ότι επίτροπος, ε, η νέα Επιτροπός Υγείας ήρθε στην Επιτροπή μας και μας υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτρέψει το θέμα του κανονισμού HTA να ξεχαστεί. Δεν το βρήκα όμως ε, στις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Και δεν τολμώ καν να σας ερωτήσω τι θα κάνετε γι' αυτό, μια που δεν βρίσκεται ανάμεσα στις προτεραιότητές σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ερωτήσω ανταυτού ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνετε στο θέμα αυτό. Γίνονται συνομιλίες, υπάρχει κάποιος διάλογος μεταξύ Επιτρόπου και Συμβουλίου για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κάποιον τρόπο να προσεγγίσετε το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί φυσικά τα κρατη και θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι, μακροσκελή συζητήσει για θέματα κυριαρχίας, αλλά κυρίως πρόκειται για την πρόσβαση στα φάρμακα και την έλλειψη μιας ενιαία προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι ο μεμονωμένο ασθενής από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει τεράστια προβλήματα στην πρόσβαση. Θα σημειώνονται καθυστερήσεις στην πρόσβασή του σε φάρμακα. Και το Συμβούλιο πρέπει να κάνει κάτι, διότι βλέπουμε ότι και η επίτροπο και εμείς ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θέλουμε να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το διέξοδο. Εσείς λοιπόν πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκλαβάκ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω κι εγώ και να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της ε, Κροατικής Προεδρίας ε, φυσικά δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάποιες προτεραιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω το ότι την πρώτη εβδομάδα του έτους σημειώθηκε ρεκόρ Δωρέα και μεταμόσχευση οργάνων στην Κροατία. Έχουν υποφεληθεί πάρα πολλοί ασθενείς. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τις ε, δωρεέ και μεταμόσχευση οργάνων, η Ισπανία έχει την πρώτη θέση. Η Κροατία φυσικά είναι πολύ ψηλά και έχει πολύ καλά προγράμματα για δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης έχουμε καλά προγράμματα στην αντιμετώπιση τη έλλειψη οργάνων προ μεταμόσχευση. Χρησιμοποιούμε έναν αυστηρότατο κώδικα δεοντολογίας για δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων στην ε, Κροατία, έτσι ώστε να μπορούμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε όργανα για μεταμόσχευση, να γίνονται δωρεές και μεταμοσχεύσεις. Σύντομα θα παρουσιαστούν και προγράμματα μεταμόσχευσης ε, πνευμόνων. Θα θέλαμε λοιπόν να δοθεί έμφαση στην μεταμόσχευση οργάνων στο πλαίσιο της πολιτικής για την υγεία. Θα ήθελα βέβαια να σας ρωτήσω εάν εσείς έχετε σκοπό να δώσετε έμφαση στο πρόγραμμα της ε, Κομισιόν για τα, τις μεταμοσχεύσεις κοιτάνων και ιστών. Η υγεία είναι πλούτος, όπως λέμε, και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε καλή υγεία. Η Κροατία θα κάνει ό,τι μπορεί λοιπόν για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ευχαριστώ τον Υπουργό για αυτά τα οποία μας είπε. Όπως λέγεται στο Mission Letter της κυρίας Κυριακίδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από μια ξεκάθαρη στρατηγική για την πρόσβαση σε αποτελεσματικά φάρμακα με ε, προσβάσιμες τιμές. Μόνο βέβαια τα γενώσιμα ε, μπορεί να βοηθήσουν προς την κατάσταση αυτή σε βασικούς ε, ε, κανόνες της υγείας στην Ευρώπη. Τι σκοπεύει να κάνει λοιπόν η Κροατία, η Προεδρία η Κροατική, έτσι ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στα σωστά φάρμακα. Μήπως θα πρέπει να κάνει μια διαβούλευση ασθενών, πληρωτών, ε, ερευνητών και ιατρικών ε, εμπειρογνωμόνων. Τώρα για την καταπολέμηση του καρκίνου, για την πρόεδρο κυρία Φόντερ Λάιεν, θα υπάρξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο. Είναι σημαντικό η στρατηγική αυτή να γίνει πραγματικότητα, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, με ολιστικό τρόπο, συγκεντρώνουμε στην προσοχή μας και στον τομέα της θεραπείας αλλά και στην πρόληψη και μάλιστα ενθαρρύνοντας την έρευνα την επιστημονική που θα πρέπει να στηριχθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σκοπεύει να κάνει γι' αυτό η Κροατική Προεδρία. Ε, τέθηκαν επίσης και πολλές ερωτήσεις για το Nutri-Score. Η επιστημονική βάση του Nutri-Score είναι βασική. Είναι θεμελιώδης. Πρέπει να ενημερώνουμε τους πολίτες. Δεν θέλουμε να τους επιβάλλουμε κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει όλα να βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες. Solis. Ευχαριστώ Υπουργέ, σας καλωσορίζω. Το θέμα της ε, μεταμόσχευσης οργάνων είναι ε, βασικό στόχος. Άκουσα με ικανοποίηση αυτό που είπατε. Εμείς είμαστε υπερήφανοι στην Ισπανία διότι είμαστε πρωτοπόροι στον κόσμο στο θέμα των μεταμοσχεύσεων οργάνων. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια στην Ευρώπη και στον τομέα της δημόσιας υγείας και στον τομέα της θνησιμότητας των παιδιών και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με το βάρος των ασθενών κτλ. Επίσης πρέπει να υπάρξει σωστή ενημέρωση για τα τρόφιμα τα οποία αγοράζουν οι πολίτες και σχετικά με το farm to fork ε, θα λειτουργήσει σωστά το σύστημα αυτό το οποίο προβλέπεται με τη σωστή ετικετοθεσία και σήμανση των προϊόντων έτσι ώστε να είναι διαφανής η προέλευσή τους και τα, και τα χαρακτηριστικά τους. Και θα ήθελα να μάθω επίσης Dos objetivos, mejorar la disponibilidad de tecnologías de la salud y hacer un uso más eficiente de los recursos. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και επιμέρους ασθένειες ε, για τις οποίες ε, θα πρέπει να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις αν έχουν πραγματικά ξεκινήσει. For the EPP, um, Novak. Novak.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 χούμανο Τι Με ένα τεχνικό πρόβλημα. Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να διευμηνεύσουμε. No, no translation. Translation problem in English. Dutch. What? Υπήρχε ένα τεχνικό θέμα, τώρα έχει διορθωθεί. Should they begin again? It was a technical. problem. If you could start again, even shortly. Okay. Yeah. Želim uspešno predsedovanje, gospod minister. Govorili ste o Ευχαριστώ, Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχηθώ ότι καλύτερο στην Προεδρία σας. Στα θέματα των, μεταναστε... των μεταμοσχεύσεων, ιδιαίτερα στα νεφρά, και η δική μου χώρα, η Σλοβενία, έχει πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν απορίες, υπάρχουν δισταγμοί σχετικά με τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται, υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις, πώς μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες να δείξουν εμπιστοσύνη στο σύστημα. Μιλήσατε επίσης και για τη γύρανση του πληθυσμού Έχουμε συζητήσει επί μακρόν ε, το θέμα της φροντίδας των ηλικιωμένων και υπάρχει επίσης και πάρα πολύ μεγάλη πίεση σχετικά με το θέμα της ευθανασίας. Ε, σε κάποιες χώρες υπάρχουν τέτοιες προβλέψεις, αλλά και εκεί η ενημέρωση δεν είναι πλήρης και οι φοβίες ε, που υπάρχουν για τις καταχρήσεις είναι παρούσες. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον της ε, μεθόδου αυτής. Αλλά στις χώρες όπου είναι νόμιμη ε, μπορούμε να έχουμε από πλευρά των ευρωπαϊκών οργάνων μια ορθότερη ενημέρωση. Η τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Ζήλη ε, κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για το κόστος παραγωγής ε, των ε, φαρμάκων. Πολλές χώρες έχουν οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν λοιπόν να πληρώσουν τις υψηλές τιμές των φαρμάκων για ορισμένες θεραπείες. Αυτό οδηγείται σε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, ε, τους ε, προνομιούχους και τους ε, μη προνομιούχους. Υπάρχουν ορισμένοι λοιπόν που περιμένουν πάρα πολύ καιρό για να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω εσείς τι προτίθεστε να κάνετε λοιπόν για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, για να ε, εξαλειφθούν αυτές οι κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της πρόσβασης στα φάρμακα και του κόστου, και του της παραγωγής. Ευχαριστώ. poštovane Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ και πάλι για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες, όσο μπορώ καλύτερα και όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις εδώ. Αν υπήρχαν, θα τις είχαμε δώσει τις ε, λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ιδίω ό,τι αφορά αυτού τους δύο φακέλου ε, όπως είναι η πρόσβαση στην περίθαλψη. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά. Φυσικά υπάρχει μεγάλος αντίκτυπος ε, ε, της φαρμακευτική βιομηχανία που θέλει να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερα κέρδη. Και βλέπουμε συχνά κάποιες χώρες να γίνονται πιο εσωστρεφείς. Και έτσι δεν είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί αντιμέτωποι με την ε, βιομηχανία του φαρμάκου. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν τα έχουμε καταφέρει ενδεχομένω, αλλά μπορεί να τα πετύχουμε στο μέλλον. Γι' αυτό και προσπαθούμε να τα συζητούμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αν καταφέρουμε να υπάρξει συμβιβασμό ε, και συνένεση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουμε κάνει και σε τόσο άλλα ζητήματα εξάλλου, θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση στην τεχνολογία, πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα τονίζουμε ξανά και ξανά κατά τη διάρκεια τη προεδρία μα, σε μια σειρά προγραμμάτων και μέτρων για παράδειγμα, υπάρχουν συγκεκριμένα έργα τα οποία υλοποιούνται ε, σε συγκεκριμένες ομάδες χωρών, αλλά αυτό μπορεί να διευρυνθεί και να επεκταθεί. Τώρα υπάρχουν ε, πράγματα τα οποία θα αποτελέσουν πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των σημαντικών δυνατών με παράλληλη τήρηση των προτύπων. Ξέρουμε ότι στον κλάδο της ιατρικής συχνά οι φαρμακευτικές ε, προωθούν συγκεκριμένα φάρμακα. Το γνωρίζει ο κόσμος και ξαφνικά μετά από 2-3 χρόνια εξαφανίζεται το φάρμακο. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι έχουν έτσι σπαταληθεί δισεκατομμύρια. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και μία ενημέρωση και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Να γνωρίζουν δηλαδή όλοι πόσο διαθέσιμο θα είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν. Να ακούσουμε λοιπόν τις φορές των ειδικών, των επιστημόνων και να ξέρουμε ότι η επιθυμία για ένα φάρμακο δεν είναι μόνο η επιθυμία για τη θεραπεία. Χρειάζεται διάλογος και με τον κλάδο και με όλους. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο να επιτευχθεί. Πρέπει να βρεθεί ισορροπία μεταξύ των αναγκών και των επιθυμιών των ασθενών και της άλλης πλευράς που προσπαθεί να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερα κέρδη. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα κάνουμε λοιπόν όσο γίνεται περισσότερες ε, συναντήσεις για να έχουμε πλήρη εικόνα από πλευράς ειδικών και επιστημόνων για τα φάρμακα του μέλλοντος, τις θεραπείες του μέλλοντος, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά γίνονται με σαφή κριτήρια. Και όταν θα είναι απαραίτητο, το φάρμακο θα μπορεί να χορηγηθεί στον ε, ασθενή. Και όλα αυτά με μια προσιτή τιμή, για να μπορεί να καλυφθεί το κόστος. Κάποιες φορές η θεραπεία για έναν ασθενή μπορεί να κοστίζει εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε την θεραπεία σε όλους. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις αναπτυγμένες με τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες και στην περίθαλψη, να αποφεύγουμε τα λαϊκιστικά μοντέλα και πρότυπα. Και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην περίθαλψη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. για τους καρκινοπαθείς, εμείς αγωνιζόμαστε ε, προκειμένου αυτοί οι ασθενείς να λάβουν την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και παρακολούθηση μετά τη θεραπεία τους για να μην ε, επανέλθει η νόσος. Γιατί στο 35% των περιστατικών επανέρχεται η νόσος ή άλλη παρεφερής νόσος. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς και από ψυχολογικής άποψης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι παίρνει από το χέρι μας για να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ε, νόσους. Και πάλι θεωρούμε ότι το καλύτερο εδώ είναι να συγκεράσουμε τις ε, δυνάμεις μας και τις προσπαθίες μας. Κάτι άλλο που ήθελα να πω. Μιλήσαμε για τη μεταμόσχευση. Μου δόθηκε εντύπωση ότι είναι σαν να αναφερόμαστε μόνο στην ε, μεταμόσχευση ε, οργάνων, αλλά πλέον στην ιατρική μιλούμε πάρα πολύ και για την μεταμόσχευση κυτάρων και ιστών. Και εδώ σημειώνονται απίστευτες εξελίξεις. Έχουμε ε, κύτταρα της σπονδυλικής ε, στήλης ε, ή και βλαστοκύτταρα που μπορούν να μεταμοσχευθούν, πρέπει να ξέρουμε πόση ποσότητα διατίθεται προς μεταμόσχευση. Να ξέρουν λοιπόν πόσα τέτοια κύτταρα και ιστούς έχουμε για να γίνει και σωστά διαδικασία. υπήρξε μια αναφορά στην έρευνα. Βλέπουμε όμως ότι σε μεγάλο βαθμό το μονοπόλιο της έρευνας το κατέχουν οι φαρμακευτικές, οι οποίες επενδύουν πολλά στην έρευνα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για το κομμάτι της ε, για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε όσο γίνεται περισσότερα κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό στην έρευνα. Είναι ένας ε, σημαντικός τρόπος για να προωθήσουμε βράχη και μακροπρόθεσμα την ευημερία. Βέβαια, δεν είμαστε εμεί εκείνοι που αποφασίζουν ε, τη μορφή που θα λάβει ο προπολογισμό. Θα ασκήσουμε όμω πιέσει, γιατί η έρευνα μπορεί πραγματικά να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο. Συνάδελφο από τη Σλοβενία μίλησε για, ε, για το πώς μπορούμε να βρούμε περισσότερους ε, δότες. Είναι δύσκολο. Έχουμε όμως πλέον κάποια εμπειρία σε σχέση με πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε τις προσπαθίες μας. Στο δικό μας σύστημα, τι κάναμε για τους ε, χρόνια νοσούντες που ξέραμε ότι τελικά θα κατέληγαν, είχαμε μία ομάδα αναισθησιολόγων, ψυχολόγων, που μιλούσαν με τους ε, συγγενείς και υπήρχε μεγάλη στήριξη. Διοργανώναμε συναντήσεις και ακόμα και με δημοσιογράφους για να αναδείξουμε τη θετική πλευρά της μεταμόσχευσης, γιατί να γίνει κάποιος δότης. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από βήματα και μέτρα που μπορούμε να μοιραστούμε με άλλες χώρες ε, σε αυτή τη συζήτηση. Και θεωρώ ότι με λίγη προσπάθεια μπορούν να βελτιωθούν ε, τα στατιστικά. Τα πρώτα πέντε χρόνια τριπλασιάστηκε ο αριθμό των μεταμοσχεύσεων. Για την ευθανασία που έδειξε κάποιο προηγουμένω. Κάποιες φορές η ιατρική δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ό,τι και να κάνουμε, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε πάντα να βοηθήσουμε όλους τους ασθενείς. Τώρα το αν μπορεί κάποιος να αποφασίσει πότε θα πρέπει να δώσουμε τέλος στη ζωή κάποιου, αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση, ιδίως αν υπάρχουν και ε, περιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρχει και δόλος. Και εδώ βέβαια έχουμε χώρες ε, που έχουν ε, θεσμοθετήσει την ευθανασία με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Μπορούμε να εξετάσουμε και αυτά τα παραδείγματα. Εγώ είμαι κατά της ευθανασίας, γιατί δεν θεωρώ ότι έχουμε το δικαίωμα να βοηθήσουμε κάποιον ε, να δώσει τέλος στη ζωή του. Αλλά επειδή έχουμε αυτό το ανοιχτό πνεύμα που προανέφερα, είμαστε διεθυμένοι να συζητήσουμε οποιοδήποτε ζήτημα Σίγουρα θα υπάρξουν και διαφωνίες. Γιατί εντάξει, άλλοι λένε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που υποφέρουν πραγματικά. Δεν αντέχουν ε, τον πόνο και μήπως εκεί θα ήταν καλύτερο. Πρέπει να το συζητήσουμε. Απλώς πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε περίπτωση κατάχρησης. Και τέλος, ε, για την ίση πρόσβαση ε, στο φάρμακο. Κατά τη διάρκεια της κρατικής προεδρίας θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε όλοι μαζί από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρχει συνένεση στην προσέγγιση. Δεν θέλουμε η κάθε χώρα ξεχωριστά να χειριστεί το ζήτημα. Θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και όσο γίνεται πιο φτηνές λύσεις. Thank you very Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ακούσαμε αυτά που είπατε, ακούσατε και από πλευρά μα πολλές παρατηρήσεις και συγκεκριμένες ερωτήσει στους τομείς του οποίους περιμένουμε από την Προεδρία να μα βοηθήσει να προχωρήσουμε. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, καλή τύχη στις προσπάθειές σας. So we are going, we are five minutes ahead, but I think. Λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μπροστά μας. I will start. We will, we will resume the, the, the NV meeting and we will start with the adoption of the agenda. Υιοθέτηση των πρακτικών. Ε, συγγνώμη, ημερήσια διάταξης. Δεκτή. Λοιπόν, πέρα από τους ε, συνήθεις υπόπτους, έχουμε τις γλώσσες ε, ηλεκτρονικά, μπορείτε να τη διαβάσετε. Κάτι που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η ενακτήρια συνεδρίαση της ομάδας για τον, εργασίας για την υγεία στις 12.30 αύριο. Θα συμπροεδρεύουν οι συμπρόεδροι και θα μας παρουσιάσουν δύο εμπειρογνώμονες τις πρόσφατες μελέτες τους. Οφέλη της πολιτικής της κοινοτική στον τομέα της υγείας και πολιτικές υγείας σημερινή κατάσταση. Ε, σας καλούμε να συμμετέχετε όλους. Και το δεύτερο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι η ημέρα του καρκίνου, 4 Φεβρουαρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με την Αρμόδια Επίτροπο θα ε, ανακοινώσει το μελλοντικό ε, της εξελίξεις για το μελλοντικό πρόγραμμα καταπολέμησης του καρκίνου στην Ευρώπη. Λοιπόν, για αύριο και για τις 4 Φεβρουαρίου τα δύο αυτά συμβάντα. Έχουμε και νέους συναδέλφους στη Γραμματεία Κανονικά δεν μιλάω εγώ. Η κυρία Κουζεύσκα είναι η νέα βοηθός μας, νέα συνεργάτης. Και η Μπρυφ, Αγγέλικα Μπρυφ, που ήταν εδώ αλλά έχει επανέλθει. <laughs> That's a welcome. Uh, thank you, Bess. <laughs> okay, so uh, Okay, so the next item is the uh, reporting back on uh, trilogues. So... Λοιπόν, τριμερείς διάλογοι και ψηφοφορίες που έρχονται σύντομα για το λεγόμενο ταξόνομη. Έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία στις 16 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, πολύ κοντά στις θέσεις του Κοινοβουλίου σε αρκετούς τομείς και θα ψηφίσουμε μαζί με την ΕΚΟΝ. Ξέρετε ότι είναι μεικτό το κείμενο. Στις 23, στις 9 το πρωί, η ημέρα πέμπτη. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να είστε παρόντες για να ψηφίσετε την Πέμπτη το πρωί. Ήταν δύσκολη η πορεία μέχρι σήμερα. Γι' αυτό παρακαλώ την κοινή αυτή προσπάθεια και η συνάντηση δεν θα κρατήσει πάνω από 15 λεπτά. Είναι κοινή μαζί με την άλλη αρμόδια επιτροπή. 23 του μηνός. Η δεύτερη ψηφοφορία για την τελική συμφωνία είναι η κατανάλωση, η ποιότητα του πόσιμου νερού μάλλον, βελτίωση της πρόσβασης σε καθαρό νερό, το δικαίωμα στην ίδρυυση. Για πρώτη φορά έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε το θέμα των νέων μορφών μόλυνσης από ενδοκρινικούς διαταράκτες και μικροπλαστικά. Την επόμενη εβδομάδα και αύριο θα ψηφίσουμε και τον τελευταία συμφωνία του ημερούς διαλόγου για τις ελάχιστες απαιτήσει. θέματα στα οποία συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου. Κλείσαμε αυτούς τους τρεις φακέλους με τη Φιλανδική Προεδρία. Ήταν μια καλή προσπάθεια και πρέπει να το αναφέρουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Συστάσεις των συντονιστών της 9ης Ιανουαρίου. Έχουν ήδη διανεμηθεί ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ. Περνάμε στο επόμενο. It's the, the big one for this afternoon που είναι το βασικό θέμα για σήμερα το απόγευμα. Ο εισηγητής είναι εδώ και οι διαπραγματευτές είναι παρόντες, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η Εστέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, ο φάκελος έχει να κάνει με τους ε, συντελεστές ε, συμμόρφωσης στις ε, δοκιμές ε, εκπομπών ε, σε πραγματικές συνθήκες. Βλέπουμε ότι δεν θέλουμε να αυξήσουμε τα επίπεδα NOx. Έχουμε τα 18 μιλιγκράμμ για αυτά τα φορτηγά και με ένα συγκεκριμένο ε, όριο σφάλματο εξαιτία ορισμένων τεχνικών αβεβαιοτήτων και στατιστικών αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τον εξοπλισμό. Θα μιλήσω αργότερα για την τυποποίηση του εξοπλισμού, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια, καλό είναι να γίνει αυτή η συζήτηση ευρύτερα, όχι μόνο για το όριο, αλλά γενικά και για το ίδιο το όριο σε ό,τι αφορά τα <clears throat> διοξίδια του αζότου που έχει να κάνει με την πρόταση Euro 7, Euro 6. Ζητούμε από την Επιτροπή να καταθέσει προτάσεις ε, στο πρώτο εξάμεινο του 2021. Από νομικής άποψης πρέπει να είμαστε ορθοί. Πρόκειται για μία διόρθωση μετά από την ε, δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Καθώς η Επιτροπή είχε προσπαθήσει να εισαγάγει ή να αποκαταστήσει ε, κάποιους συντελεστές συμμόρφωσης ε, που είχε για το 2016. Ξέρω ότι υπάρχει έφεση, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι. Να εργαστούμε από κοινού βάσει της ε, συναπόφασης τελικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βασιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα και για τον τελικό συντελεστή συμμόρφωσης από το 1,5 τελικά πήγαμε στο 1,43 βάσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου που αντικατόπτριζαν βελτίωση στην ακρίβεια των PEMS, αυτών των φορητών μετρητών. Μπορούμε να κάνουμε εκ νέου αναθεώρηση προς τα κάτω και πάλι βάσει στοιχείων του JRC. Η έκθεση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει τους συντελεστές συμμόρφωσης, να τους αναθεωρεί κάθε χρόνο, βάσει της ενδεχόμενης βελτίωσης ε, των αποτελεσμάτων των μετρητών και βεβαίως ε, θα ακούσουμε τα χαράς ε, και τους σκιώδης. Δύο ερωτήματα όμως θα θέλω να απευθύνω, Πρόεδρε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δημοσίευση της έκθεσης του JRC είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, αλλά τώρα βλέπω ότι αναβάλλεται για τον Φεβρουάριο. με βάση τι πληροφορίες που έχω λάβει, ε, αποφάσισαν να προσθέσουν πληροφορίες στην ανάλυση τους, το οποίο είναι αρκετά ασαφέ. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιες είναι αυτές οι επιπρόσθετες πληροφορίες και τελικά όντω το Φεβρουάριο θα λάβουμε την έκθεση. Γιατί όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας ε, ε, σκεφτόμαστε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή το JRC να έχει το 1,32 ως ε, μέγιστο συντελεστή συμμόρφωσης, και είναι σημαντικό για την ομάδα διαπραγμάτευση ε, να γνωρίζει με σιγουριά τι γίνεται. Μπορεί να αναθεωρηθεί δηλαδή αυτό το νούμερο. Τέλος πάντων, ξέρετε εσείς γιατί πρέπει να προσθεθούν και άλλες πληροφορίες στην ανάλυση. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, για την τυποποίηση των PEMS. Δεν έχει λήξει ακόμα το θέμα, αλλά δεν έχουμε λάβει απάντηση για το πότε θα γίνει αυτό και είναι σημαντικό τα PEMS να χρησιμοποιούν τις ε, καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές στην αγορά. Ξέρετε και ο Σεν ασχολείται με αυτό, αλλά μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι γίνεται η θητεία αυτή, η εντολή μάλλον ε, ε, ισχύει ακόμα, είναι ακόμα κατάλληλη, πρέπει να επικαιροποιηθεί, τι μπορεί να μας πει. γιατί σε αυτά τα δύο δεν υπάρχει ακόμα αρκετή σαφήνεια για να μπορέσει να εργαστεί και η ομάδα διαπραγματεύση. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω και τι υπόλοιπε ομάδε. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο στη συνέχεια. Και επειδή δεν προβλέπετε ακόμα, αλλά και επειδή δεν έχουν φτάσει, λέει ο πρόεδρος. Α, έχετε φτάσει, εντάξει. Καλύτερα όμως να απαντήσουν ε, στο τέλος. Ωραία. Η κυρία Νταλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση χωρίς να έχουμε κατά νου το σκάνδαλο Dieselgate, τις προεκτάσεις του, την ε, σχετική επιτροπή στο Κοινοβούλιο και τις συστάσεις γιατί η ομάδα Άμυση είπε ότι ο στελεστής θα πρέπει να μειωθεί στο 1 και εδώ είχαμε συμφωνημένη προσέγγιση και από το Κοινοβούλιο. Τώρα ξαφνικά έχουμε όλη αυτή την δημιουργική προέλαση με άλλους συντελεστέ, με άλλα ονόματα. Ε, ήταν παραθυράκι, είναι παραθυράκι, ό,τι όνομα και να το δώσουμε παραθυράκι θα μείνει. Γιατί έχουμε συγκεκριμένους συντελεστέ. Το 2,1 και το 1,5 και εκείνους από τις δοκιμές ZRT επιτρέπουν στα οχήματα να εκπέμπουν 168 ένα χιλιόμετρο και 123 νόξ. Πολύ πάνω από τα 8 μιλιγκράμμα χιλιόμετρα υπό τους κανόνες του ε, Euro 6. Όπως έχουν επιβεβαιώσει πολλοί εμπειρογνώμονες, δεν ξέρουμε κατά πόσο πρέπει να συμπεριλάβουμε οποιοδήποτε συντελεστή συμμόρφωση στη διαδικασία RDT. Γιατί και πάλι υπάρχει πλήρης διάσταση με διάφορες ανεξάρτητες δοκιμές. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα οχήματα Euro 6 καθιστούν εφικτό και προσιτό οικονομικά να πετύχουμε συντελεστές συμμόρφωσης κάτω από το 1,5 και πολύ κάτω από τα 80 mg ένα χιλιόμετρο. Η συντελεστή συμμόρφωση ή οποιαδήποτε απόκληση από, τα, τον κανόνα των 80 mg ένα χιλιόμετρο στα NOx δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πια. Απλώ επιτρέπει την συνέχιση τη χρήση λιγότερο αποτελεσματικών και αποδοτικών τεχνολογιών. Η εφαρμογή λοιπόν συντελεστή συμμόρφωση ή ορίου σφάλματο ε, αποτελεί παρέκκληση από τα εφαρμοστέα όρια. Δηλαδή, τίθεται, υλοποιείται ένα ε, και επιβάλλεται ένα όριο από τη μία και από την άλλη έχουμε το παραθυράκι του. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο προηγούμενο. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν νομοθετική προσέγγιση. Μάλλον δεν, δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια νομοθετική πρόταση. Ο συντελεστή συμμόρφωση που αναφέρει η συγγήτρια η πρώτη μάλλον που αναφέρθηκε δεν ε, είναι φιλόδοξη. Τα 80 μιλιγκράμμα χιλιόμετρο είχαν υιοθετηθεί πριν από 12 χρόνια και η αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει ότι αυτά τα δεδομένα ε, έχουν από την άλλη οχήματα που μπαίνουν στην αγορά χωρίς καμία ανάγκη για ευελιξία σε ό,τι αφορά το συντελεστή και το όριο σφάλματος. Δεν γίνεται λοιπόν αυτά τα όρια που έχουν τεθεί στα 80 χιλιόμετρα να είναι αυξημένα σε σχέση με τα ε, οχήματα diesel που είναι 60 και είναι ψηλότερα στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Δεν υπάρχει λόγος να επιτρέπουμε σε μία τεχνολογία να ρηπαίνει περισσότερο από ό,τι άλλες και να δίνουμε στα diesel οχήματα ε, τη δυνατότητα να ρηπαίνουν περισσότερο οι κατασκευαστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες αντί να ποντάρουν ε, σε έναν συντελεστή συμμόρφωσης που τους επιτρέπει να εκπέμπουν ε, υψηλότερα. Υπάρχουν ε, διαθέσιμες και προσιτές τεχνολογίες για την αυτοκινητοβιομηχανία και θέλουμε οι, ακριβώς αυτές τις τεχνολογίες να εφαρμόσουν. Επομένω, η πρόταση τη Κομισιόν καθώ και η πρόταση τη εισηγήτρια του ΕΛΚ δεν θεωρούμε ότι μπορεί να μα έχει μας δώσει επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα Renew, η Σουζάννα Σόλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για την παρουσίαση τη έκθεσης. Συμφωνώ με το περιεχόμενο της έκθεσης σε γενικές γραμμές αλλά πρέπει να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι αν θέλουμε πράγματι να μειωθούν οι εκπομπές. Διότι πρόκειται για θέμα υγείας. Υπάρχουν ε, εκατοντάδες ε, πρόοροι θάνατοι ακριβώς από αυτά τα αίτια και στο πλαίσιο του Green Deal χρειάζεται περισσότερη φιλοδοξία. Θα επιμείνω λοιπόν στη φιλοδοξία αυτή πέρα από το περιεχόμενο της πρότασης του Euro 6. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες εκπομπές από τα οχήματα. Και χρειάζεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία ήταν ο Ιούνιος του 2021 μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στους παράγοντες συμμόρφωσης όπως ήταν στην αρχική πρόταση και να γίνει διαχωρισμός ε, ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Να αναλάβει τις ευθύνες της η αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει εκπομπές στα 60 μιλιγκράμμα ανά χιλιόμετρο. Επίσης, Όλα τα οχήματα από 1η Πρώτου 2020 έχουν 0,3% ποσοστό σφάλματος για τα όργανα μέτρησης των εκπομπών. Εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε την δυνατότητα αναθεώρησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μέσω πράξεων εξουσιοδότηση Και να πω επίσης ότι λάβαμε την έκθεση της Επιτροπής ε, ένα μήνα πριν ε, σχεδόν και είδαμε τότε για αυτή τη μείωση του για το, στο 0,3% Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω πως ε, θα πρέπει να μας ενημερώσει για τα νέα στοιχεία που εισήγαγε στην πρόταση. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος ακόμα περισσότερο. Όπως είπε τώρα η συγγήτρια, η τυποποίηση είναι ακόμα ένα θέμα, η τυποποίηση των ε, συστημάτων μέτρησης. Υπάρχουν διάφορα PEMS αυτή τη στιγμή στην αγορά και οι μετρήσεις διαφέρουν ε, αντίστοιχα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε έτσι ώστε να χρησιμοποιείται πάντα η πιο καινούργια τεχνολογία μέτρησης και να υπάρχουν οι κατάλληλες πιστοποιήσεις. Χωρίς αυτές τις πιστοποιήσεις ε, δεν θα καταφέρουμε να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος. Πρέπει λοιπόν αυτά τα PEMS να είναι πιστοποιημένα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ε, μέγιστη δυνατή ποιότητα. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μάθω από την Επιτροπή πού βρίσκεται ως προς αυτό. Έπειτα, συμφωνώ με την εισαγωγή του παράγοντα συμμόρφωσης. Ε, δεν είναι η καλύτερη λύση, όμως είναι κάτι που έχει εγκριθεί δημοκρατικά το 2016. Και υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ε, που πρέπει να, και πρέπει να τηρούν οι κατασκευαστέ από το 2018 και μετά. Βλέπουμε τώρα την απόφαση του δικαστηρίου για ε, αναδιαμόρφωση των παραγόντων ε, συμμόρφωσης, ε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πρώτα να ε, εγκρίνει τη διαδικασία επιτροπολογίας. Όμως αυτό θα μας ξαναφέρει στην αρχική διαδικασία και όλο αυτό προσδίδει μια βεβαιότητα που είναι το τελευταίο που χρειάζεται η αυτοκινητοβιομηχανία. Χρειάζονται μήνες και μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Και όπως είπε και η κυρία Ντάλη, το 86% των οχημάτων έχουν όριο 8 μιλιγκράμμα ανά χιλιόμετρο. Είναι πολύ θετικό λοιπόν ε, ότι βλέπουμε να πιάνουν τόπο τα μέτρα, όμως τι γίνεται με τα οχήματα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης τύπου. Ξέρετε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το ποσοστό μη συμμόρφωσης της θέσης εργασίας. Η βιομηχανία χρειάζεται ασφάλεια για να λειτουργήσει σωστά και χρειάζεται ταχύτητα λοιπόν έτσι ώστε να ε, αλλάξουν αυτοί οι παράγοντες συμμόρφωσης. Αυτό λοιπόν σας ζητώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπάσα Έκχουτ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Μου φαίνεται πως επαναλαμβάνεται η συζήτηση. Τα ίδια ακούμε τώρα, τα ίδια ακούσαμε και κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά τη στο σχέδιο έκθεση, όμω μη σα εκπλήξει η διαφωνία μου με εκείνη. Είναι θέμα συνέπεια. Τώρα νομίζω πω ε, χρειάζεται να απαντήσω στον σκιώδη εισηγητή από το Renew, γιατί μου φαίνεται πω έχουν γίνει κάποιε παρεξηγήσει. Μα είπατε καταρχά ότι το 2016 εγκρίθηκε δημοκρατικά αυτό το μέτρο. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι από το 2007 υπάρχει το όριο των 80 μιλιγκράμμ ανά χιλιόμετρο. Μικρογραμμαρίων. Από το 2007 λοιπόν είναι γνωστό στην αυτοκινητοβιομηχανία ότι υπάρχει αυτό το όριο των 80 μικρογραμμαρίων και κατάφεραν να επινοήσουν ένα σωρό κόλπα για να το προσπεράσουν και αυτό μας οδήγησε στο σκάνδαλο Dieselgate. Έπειτα τι έγινε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε μέσω πράξεων εξουσιοδότηση να αλλάξει την ε, νομοθεσία. Εμείς ε, γύραμε αντιρρήσεις, οι πράσινοι, οι τότε Άλντε, οι φιλελεύθεροι, οι Γκουε, και οι σοσιαλιστέ όμω χάσαμε στην ψηφοφορία, διότι για να γίνει μια ένσταση σε μια πράξη κατά εξουσιοδότηση χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Και για να αλλάξει αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη συνήθινη νομοθετική διαδικασία και όχι μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Το δικαστήριο πώ αποφάσισε. Αποφάσισε ότι αυτέ οι αλλαγέ δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο με τη συνήθινη νομοθετική διαδικασία και όχι με πράξη κατά εξουσιοδότηση. Είναι θέμα συνέπεια λοιπόν να ακολουθήσουμε τη συνθηνομοθετική διαδικασία. Μπορείς βέβαια στην πορεία να αλλάξεις άποψη και να πεις ότι ας πούμε εντάξει μπορούν να εισαχθούν παράγοντες συμμόρφωση σύμφωνα με τα πρότυπα του 2007, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Διότι ας μιλήσουμε ειλικρινά. Ήδη από το 2007 υπάρχουν κάποια πρότυπα των 80 μικρογραμμαρίων. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε αβεβαιότητα με τον αλλάζουμε τον παράγοντα συμμόρφωσης ε, στην ουσία αποδυναμώνοντας την αρχική πρόταση του 2007. Και θα δημιουργήσουμε προηγούμενο ότι δηλαδή από εδώ και στο εξή οποιοδήποτε όριο θέτουμε θα μπορεί να αλλάξει μέσω αυτού αυτών των αβέβαιων παραγόντων και λαγών στη συνέχεια. Φανταστείτε ότι να γινόταν αυτό στα όρια ταχύτητας. Δεν επιτρέπεται αβεβαιότητα στα όρια ταχύτητας. Τι θα λέμε, εντάξει το όριο ταχύτητας είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα, πολλαπλασιάζουμε με 1,4 για το περιθώριο σφάλματος, έτσι δημιουργούμε αβεβαιότητα ασάφεια και απέχουμε πολύ από αυτά που έχουν εγκριθεί δημοκρατικά, όπως είπατε εσείς. Και αναμένω η νέα σύνθεση της ε, ομάδας Renew να έρθει στο πλευρό μας και να μην υποχωρήσει, να μην αποδυναμώσει τα πρότυπα από την άλλη λέγοντας ναι εντάξει θέλουμε να έχουμε ένα φιλόδοξο Euro 7. Πρέπει τώρα να αλλάξουν αυτά, πρέπει τώρα να δείξουμε τη φιλοδοξία μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παροτρύνω όλους σας να μην επιτρέψετε μια τέτοια αποδυνάμωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εδώ η Σίλβια Λίμερ εκ μέρους του ID. Για την ομάδα ECR η κυρία Ζαϊόσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά η παρουσίασή σας. Εμείς όμως θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή, με την εισηγήτρια μάλλον, αν και αυτό θα σας απογοητεύσει. Νομίζω ότι εμένει σε συγκεκριμένες θέσεις κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλει η βιομηχανία να έχει μια κάποια νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Η συγχύτρια οργάνωσε μια συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον JRC. Και αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δυστυχώς παραμένουν αναπάντητα. Ε, δημιουργούνται θέματα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο JRC, ε, στο κέντρο. Πολλά προγράμματα δεν έχουν ολοκληρωθεί και μιλάμε για τεχνολογικούς τομείς τους οποίους δεν υπάρχουν περιθώρια για ατέλειες. Ελπίζω λοιπόν τα πράγματα να μετά τις εξηγήσει και τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί να βελτιωθούν. Γίνονται και νέες προτάσεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 σαν παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέσα τα οποία είναι τόσο συγκεκριμένα, τόσο λεπτομερή που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις μικρομεσαίες που θα παίρνουν μέρος. Οι μικρομεσαίες μπορεί να απομακρυνθούν με τον τρόπο αυτό από την αγορά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κονιέτσκα από την Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Σας είπα την άποψή μου γενικότερα, θα είμαι πολύ σύντομη. Η δισταγμή της εισηγήτριας, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει κάποια στοιχεία βεβαιότητας, είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας πει με ξεκάθαρο τρόπο πότε θα είναι διαθέσιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πότε θα γίνουν τα επόμενα βήματα. Ε, πριν μιλήσει ο πράσινος συνάδελφος, ο συνάδελφος από την ομάδα των Πρασίνων, είχαμε περιοριστεί στα δεδομένα. Μετά την παρέμβασή του τα πράγματα έγιναν κάπως πιο ασαφή. Πάντως πιστεύω ότι λόγω ακριβώς της έλλειψης νομικής βεβαιότητας σχετικά με το ποια θα είναι τα ανώτατα όρια και περιμένουμε την εφετική διαδικασία και ταυτόχρονα λόγω της σύντομης περίοδου για τη συμπληρωματικής τροπολόγησης και λόγω του ότι ε, δεν έχουμε ακόμα την έκθεση του Κοινού Κέντρου, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω ότι θα μπούμε σε λεπτομέρειες αντικειμενικά, ψύχρεμα ε, και μη κομματικά θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν εδώ ε, έχουμε έρθει για να λειτουργούμε συναισθηματικά και μόνο και να μην σεβόμεθα τη δική μας νομοθεσία. Γιατί σε ένα χρόνο θα έχουμε να κάνουμε με μια νέα αναθεώρηση και τότε θα έχουμε ίσως κάποια δεδομένα πολύ συγκεκριμένα. Αλλά το να κάνουμε τη συζήτηση αυτή τώρα, ακριβώς σε επισυναισθηματικής ε, ε, βάσεως ε, δεν θα ήταν υπεύθυνο και θα οδηγούσε φοβάμαι σε απαράδεκτες καταστάσεις. Θα βάλουμε στο χαρτί δηλαδή κάποια στοιχεία χωρίς επιστημονική βάση που θα δημιουργήσουν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά τα οποία θα λύσουν. Και η αναθεώρηση η οποία υποχρεωτικά θα ακολουθήσει σε 12 μήνες θα οδηγήσει σε καταστάσεις αδόκιμες θα πρέπει να φανούμε ιδιαίτερα επίοικείς και ε, να διορθώσουμε τους εαυτούς μας. Ας είμαστε λογικοί, ας είμαστε ορθολογικοί, ας περιμένουμε τα συμπεράσματα του κοινού κέντρου και να περιμένουμε ακριβώς την σωστή αναθεώρηση σε ένα χρόνο. Αυτό που είπε ο Μπάς, ότι δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, δεν είναι αλήθεια. Υπήρχαν νομικέ ρυθμίσεις οι οποίες ε, εμένα δεν μου άρεσαν αλλά υπήρχαν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε λοιπόν την αλήθεια. Θα πρέπει να σεβαστούμε την νομοθεσία η οποία είναι ενισχύ. Αυτή πρέπει να είναι η βασική μας, αν θέλετε, ε, δραστηριότητα και δεν θα πρέπει με μη καρποφόρο τρόπο να ξοδεύουμε τον συναισθηματικό μας κόσμο χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς συγκεκριμένα γεγονότα. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με το Catch Τρία αιτήματα. Τέσσερα. Καλώς. Εύη, μία εγγεγραμμένη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη περίοδο εξεφράστη επανειλημμένα εναντίον αυτών των παραγόντων συμβατότητας που δημιουργούν προβλήματα. Ήδη από το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τα ανώτατα όρια των ΟΚΣ. Μετά ήρθε το σκάνδαλο του Dieselgate πολλά οχήματα εκπέμπουν 20 φορές περισσότερο από όσο επιτρέπεται. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Τα όρια θα πρέπει να γίνονται σεβαστά σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε ένα τεχνικό εργαστήριο. Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δημιουργούν αβεβαιότητα. Ήδη από το 2011 είχε ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή και δεν απέδωσε. Για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στις αυτοκινητοβιομηχανίες, άλλαξε ο κανονισμός με τον 246 του 2016 ε, χωρίς συναπόφαση για τους παράγοντες συμβατότητας ε, που στην ουσία επιτρέπουν με νομικό τρόπο, με νόμιμο τρόπο να μην γίνονται σεβαστά κάποια όρια. Και έτσι παρενέβη το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο μας έδωσε, μας δικαίωσε και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε δικαίωμα να τροποποιήσει τη βασική πράξη για τα νόξο με μια τεχνική απόφαση. Το δικαστήριο λέει ότι η τεχνική και στατιστική αβεβαιότητα της βελτίωσης θα πρέπει να επιληθεί μέσω της βελτίωσης της αντιπροσωπευτικότητας των δειγμάτων και όχι μόνο με δειγματοληψίες προσωρινές και επιμέρους. Δέκα χρόνια χρειάστηκε αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να καθορίσει επαρκώς την πρόοδο η οποία έχει συμβεί έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, προβλήματα τέτοιου είδους. Δεν μπορώ να συμφωνήσω λοιπόν εγώ με την έκθεση αυτή η οποία θα έλεγα αδικαιολογίαν πολύ στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση αυτή και εγώ θα καταθέσω μία τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει και κάτι επιπλέον που πρέπει να καταδικάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι πρέπει επιγόντως να δράσουμε για να αποφύγουμε την νομική αβεβαιότητα έτσι ώστε να τεθεί ενισχύ η απόφαση του δικαστηρίου στις 23 Φεβρουαρίου του 20. Ψέμα. Δεν υπάρχει τίποτα το κατεπήγον. Δεν μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει καταθέσει έφεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχει αυτή τη στιγμή αναστολή των όρων τους οποίους κατά τα άλλα προτείνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι ιδιαίτερα στενάχωρη η κατάσταση και θα πρέπει σαν κοινοβούλιο ενωμένο να ζητήσει την απόρριψη της πρότασης. Thank you Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάτεμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, μπορεί να φαίνονται πολύ απλά τα πράγματα, αλλά μας έχουν εκλέξει ψηφοφόροι που πιστεύω ότι αν μας παρακολουθούν, ε, σίγουρα θα έχουν μπερδευτεί. Α, και ο Νίλς με έχει ψηφίσει. Αν δείτε το 2007, είχαμε καταλήξει σε αυτά τα πρότυπα, σε αυτούς τους κανόνες. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε αν όλοι συμφωνούν. Εφόσον όμως έχουμε συμφωνήσει, πρέπει όλοι να ακολουθούμε τους κανόνες. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Όποιος αγοράζει ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να κατανοήσει ποια είναι η κατανάλωσή του. Μπορεί κάποιο να, να του λένε από την αντιπροσωπή ότι είναι χ ε, η κατανάλωση και εκπομπέ, αλλά μετά τελικά στην πράξη να είναι διπλάσια τριπλάσια. Και μετά απεδείχθη ότι αυτό έγινε σε, σε εργαστήριο. Έγιναν αυτές οι πλαστές ε, δοκιμές με λογισμικά που προσπαθούσαν να μαγειρέψουν τα αποτελέσματα. Από αυτή την άποψη, ε, η εικόνα της αυτοκινητοβιομηχανίας φυσικά δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγμα στη συνέχεια, αντί να πούνε εντάξει τώρα πρέπει να σοβαρευτούμε και να διασφαλίσουμε ότι οι εκπομπές που αναφέρουμε είναι πραγματικές, τελικά έχουμε έναν συντελεστή συμμόρφωσης. Είχαμε το 1,5, 40%, 20%, όλα αυτά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Εμείς χρειαζόμαστε νομοθεσία που θα λέει αυτά είναι τα κριτήρια, αυτοί είναι οι κανόνες, πρέπει να πληρούνται από όλους. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Πάουλου. Αυτό ακριβώ μου έλεγαν και εμένα οι ψηφοφόροι κατά την προεκλογική εκστρατεία. Πώς γίνεται να έχουμε νομοθεσία και απλά να μην ακολουθείτε από την αυτοκινητοβιομηχανία. Πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιος άλλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το στρίξει τα δόντια και να ε, υλοποιήσει τον ε, νόμο, να τους αναγκάσει να τον ακολουθήσουν. Εγώ δεν έχω πιστεί σε σχέση με όλο αυτό το αφήγημα για την ε, ε, νομική εξασφάλιση, γιατί πρέπει να υπάρχει έκθεση που θα αποκλείει οποιαδήποτε ασυνέπεια. Οι δικοί μας καταναλωτές περιμένουν να τους δώσουμε όλες τις τιμές που έχουμε μετρήσει και με τις αβεβαιότητες που μπορούμε να υπολογίσουμε αν ξέρουμε τι κάνει ο εξοπλισμός μας και αν όλα αυτά γίνονται σε σωστά εργαστήρια και γίνονται δοκιμές για να βρούμε ακριβώς ε, τα όρια ασφάλματος που έχει ο εξοπλισμός μας. Αυτό ποτέ δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία. Όταν ο δεν μπορεί να έχει ένα σωστό εργαστήριο, τι να την κάνει την νομοθεσία. Δεν, έχει, δεν χρειάζεται καινούργια νομοθεσία. Δεν, πρέπει να, θα έπρεπε να είχαμε αποδεχθεί κανέναν συντελεστή συμμόρφωσης. Ο κύριος Κόκαλης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να μιλήσω για τα εργαστήρια. Με προβληματίζει όλη αυτή η χρήση των όρων ε, συναισθηματισμό, τρομολαγνία και ούτω καθεξής και ότι πρέπει να σταθούμε στα επιστημονικά στοιχεία. Νομίζω ότι τα εργαστήρια είναι χώροι που στερούνται συναισθημάτων, αλλά σε πραγματικές συνθήκες υπάρχουν πολλά συναισθήματα, ιδίως ό,τι αφορά τι εκπομπές NOx, που δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, έχει να κάνει με τη ρήπανση και ανθρώπινες ζωές. 374.000 πρόοροι θάνατοι κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέρη εξαιτία τη ε, ρήπανση. Χωρίς συναισθηματισμούς το λέω αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ε, χώρος ε, για συναισθηματισμούς από νομικής άποψης. Υπάρχει νομική διαδικασία που πρέπει να τηρείται. Να τηρούνται οι νόμοι λοιπόν και να μην καταφεύγουμε σε διάφορες τέτοιες ε, εφευρέσεις και επινοήσεις όπως ήταν αυτός ο συντελεστής συμμόρφωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ο κ. Στόρβαλτς. Ένα σχόλιο προς τον Μπάς περισσότερο. Για αυτά που είπε για το Ρινιού. Υπάρχει ακόμα συζήτηση. Ήδη τα συζητήσαμε προηγουμένως στην πολιτική μας ομάδα και θα τα ξανασυζητήσουμε εν ώψη της ψηφοφορίας από μία άποψη έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από τη πράσινη. Συνήθως ε, είναι ο Μπάς Άικχαουτ, εισηγητής, η για, για τα πάντα. Καλό είναι βέβαια αυτό για τον ίδιο, αλλά κάποιες φορές γίνεται λίγο μονόπλευρη η συζήτηση. Εμείς έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Αφήνουμε περιθώριο ελευθερίας στα μέλη μας και μετά κάνουμε και μια συζήτηση. Ελπίζω να εκτιμήσεις ε, την προσέγγισή μας και θα δεις τα θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή που έθεσε η Έστερ Ντελάνγκε. Έστερ, μπορείς να επαναλάβει τα δύο ερωτήματα. Βέβαια, βέβαια, κανένα πρόβλημα. Είχα μια ερώτηση για την έκδοση της ε, έκθεση σε JRC. Γιατί λοιπόν υπάρχουν ορισμένες ε, πληροφορίες που προσθέθηκαν στην ανάλυση. Ποιες είναι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες και εάν η προθεσμία του Φεβρουαρίου είναι η τελική. Αυτό επίσης που ανέφερε και το Renew είναι η τυποποίηση των PEMS. Τα PEMS δεν πρέπει να είναι οτιδήποτε, αλλά η καλύτερη δυνατή τεχνολογία με ε, εξοπλισμό ακριβίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα της ε, τυποποίησης ε, και δεν με εκπλήσει που οι απαντήσεις είναι έτσι ασαφείς. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει πού ακριβώς βρισκόμαστε και αν ε, επαρκεί η εντολή, αν χρειάζεται ανανέωση. Πότε μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο έκθεσης. Να ευχαριστήσω λοιπόν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έγκρισή σας στην πρότασή μας. Οι αλλαγές που προτείνατε θα αποσαφηνίσουν το κείμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, για την έκθεση GRC, χρειάζεται να πω ότι η αρχική μας εκτίμηση είναι ότι θα... εγκρινόταν τον Ιανουάριο μετά από τη συζήτηση όμως που είχαμε το Δεκέμβριο είδαμε πως είχαν προκύψει ορισμένες ερωτήσεις του Κοινοβουλίου για την ε, αντιπροσωπευτικότητα των ε, πληροφοριών που είχαμε και σχετικά με την ε, ποιότητα του εξοπλισμού που υπάρχει στην αγορά. Έχουμε εξετάσει λοιπόν το 75% του διαθέσιμου εξοπλισμού. Αυτό για ορισμένους από εσά δεν επαρκεί για να γίνει μια πλήρης αξιολόγηση των δυνατοτήτων των ε, διαφορών PEMS, των συστημάτων μέτρησης λοιπόν. Χρειάζεται λοιπόν σύμφωνα με ορισμένους από εσά μία μελέτη που να καλύπτει το 100% και αυτό φυσικά οδηγεί σε καθυστερήσεις. Ε, σύντομα θα έχουμε αυτή την ε, ανάλυση, αυτή την ερχόμενη εβδομάδα περίπου ή τη μεθεπόμενη. Και ο σκοπός δεν ήταν να καθυστερήσουμε, αλλά να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Περί τα τέλη Ιανουαρίου είχαμε μια αρχική εκτιμόμενη ημερομηνία για τα αποτελέσματα, όμως τώρα θα πάμε λίγες μέρες ε, πίσω, περίπου αρχές Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα πρότυπα. Στις αρχές του μήνα λάβαμε μία έκθεση από την ομάδα εργασίας που καταρτίζει τέτοια πρότυπα. Ο στόχος ήταν να εγκριθεί περί τα μέσα Μαρτίου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε περίπου 2-3 εβδομάδες καιρό για να αναλύσουμε το περιεχόμενο της έκθεσης, τα πορίσματα της ομάδας εργασίας, να δούμε τις προτάσεις με προσοχή και να αξιολογήσουμε την ποιότητα της ε, έκθεσης. Περίπου λοιπόν στα μέσα Μαρτίου αναμένουμε την έγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έψαχνα απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας τις έδωσε. Ε, να ευχαριστήσω και για τις λεπτομέρειες σχετικά με τα JRC. Ήταν κάτι που είχε ζητήσει η Επιτροπή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών. Θα δούμε τι θα καταθέσουν οι συνάδελφοι και ελπίζω να καταφέρουμε να είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία και να καταλήξουμε σε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Ναι, αλλά ξέρετε, ορισμένε φορέ κρύβει στην πολυμορφία στην ε, ενότητα. Να δούμε πώς θα τα συνδυάσουμε λοιπόν αυτά τα δύο. Μήπως θα ήταν καλύτερο να δώσουμε μια παράταση στην ε, ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα της έκθεσης JRC, να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο της έκθεσης γιατί η ημερομηνία, καταληκτική ημερομηνία για τις θα είναι πριν τη δημοσίευση της έκθεσης JRC. Καλό θα ήταν λοιπόν να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο της έκθεσης πριν καταθέσουμε τροπολογία. Νομίζω πως ε, για να διατηρηθεί αυτή η ενότητα καλό θα είναι να περιμένουμε. Καταλαβαίνω από την συζήτηση ότι τουλάχιστον δύο, ενδεχομένως και τρεις πολιτικές ομάδες, οι οποίες θα καταθέσουν ε, τροπολογίες και προτάσεις ε, και για, τον, ε, για τους παράγοντες συμμόρφωσης. Τώρα, δεν βλέπω το λόγο να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, διότι, όπως σας είπα, οι ομάδες έχουν ήδη αποφασίσει να έχουν το ένα ως παράγοντα συμμόρφωσης. Ναι, η πρόταση του Μπα σχετικά με τους παράγοντες συμμόρφωση αφορούσε την ημερομηνία. Είναι λογικό πιστεύω αυτό που λέει ο Μπάς. Τέλο πάντων, για να σας λύσω τις απορίες, η συγκήτρια θα αποφασίσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τα σχόλιά σας. Αν αλλάξετε άποψη για την διαπραγματευτική ομάδα είναι κάτι που θα το αποφασίσουν άλλοι και όχι αυτή εδώ. Η Επιτροπή. Λοιπόν, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 28 Ιανουαρίου. Ψηφίζουμε το Μάρτιο στην Επιτροπή. Δεν θα ξεκινήσουμε τώρα συζήτηση για αυτό το θέμα. Να κλείσουμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης, να το ολοκληρώσουμε και να περάσουμε στο σημείο 8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112, παράγραφοι 2 και 3 και 4 για την καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμού των χημικών προϊόντων όσον αφορά το μόλιβδο και τις ενώσεις του, PVC. Θα δώσω το λόγο ξανά στον Bass out. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτός ο φάκελος, ε, θα έλεγα, έχει ξεκινήσει ήδη ε, πολύ παλιά, από το 2000. Το 2000 ήδη συζητούσαμε ε, το θέμα της χρήσης του PVC, ε, της χρήσης ορισμένων σταθεροποιητών μέσα στη, για την κατασκευή του PVC ε, ε, that there are no safe levels that can be determined uh, by that. Ε, υπήρχε λοιπόν μια πράσινη βίβλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000 για το μόλιβο. ήδη από το 2001 είχαμε ζητήσει την απαγόρευση του μολύβδου στο PVC. Αυτό έχει ξεκινήσει λοιπόν εδώ και πάρα πολλά πολλά χρόνια. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε άλλα στο νου της και αποφάσισε ε, να προχωρήσει σε μια εθελοντική σταδιακή αποχώρηση θα έλεγα που θα ολοκληρωνόταν το 2015. Και έτσι λοιπόν ε, υποτίθεται ότι ε, από το 2015 δεν θα υπήρχε μόλιβδο στα PVC, ενώ εμείς θέλαμε να σταματήσει αμέσως, η Επιτροπή αποφάσισε διαφορετικά. Τώρα βέβαια έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, ότι αυτή η εθελοντική συμφωνία δεν αφορά τις εισαγωγές PVC. Και τώρα λοιπόν είμαστε στην περίεργη κατάσταση όπου έχει απαγορευτεί πλέον η χρήση ε, στο PVC στην Ευρώπη, αλλά έχουμε προϊόντα PVC που εισάγονται. Και γι' αυτό ακριβώς κάνει την πρόταση περιορισμού ε, χρήσης μολύβδου στο PVC. Ε, περιορισμός ο οποίος λέει όχι δεν θέλουμε ότι λέμε στην ευρωπαϊκή αγορά όχι μολύβδο αλλά εμείς μιλάμε για ένα διοικητικά επιτρεπόμενο όριο για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα, η Επιτροπή λέει καλύτερα από το τίποτα. Αλλά ταυτόχρονα εμείς επιτρέπουμε και εξαιρέσεις. Επιτρέπουμε εξαιρέσεις ε, για ανακυκλούμενο PVC. Δημιουργούμε λοιπόν μία διαφορετική, αν θέλετε, αγορά και επειδή είχαμε παρόλα αυτά πολλά προϊόντα τα τελευταία χρόνια, λέμε ότι μπορεί τα προϊόντα αυτά να χρησιμοποιηθούν εκ νέου. Στην ουσία χρησιμοποιούμε την επιχειρηματολογία της ανακύκλωσης τώρα για να επιτρέψουμε ουσιαστικά περισσότερο την παρουσία του μολύβδου στο PVC. Αυτά είναι εντελώς κατά σε αυτά τα οποία είχαμε αποφασίσει μέχρι σήμερα και οι συνάδελφοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δεν έχουν καταλήξει ακόμα και συνειδητοποιώ, Πρόεδρε, και τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας και το χρόνο που χρειάζεται. Αλλά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υιοθέτησε την προηγούμενη εβδομάδα το λεγόμενο Green Deal και μιλάει για μη τοξικά προϊόντα, για κύκλους μη τοξικών προϊόντων που το λέει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει ξεκάθαρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν θα πρέπει να επανεισαχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης. Και ακριβώς αυτό κάνουμε. Εμείς στην ουσία επιτρέπουμε μέσω της ανακύκλωσης να συνεχίσει ο μόλιβδος να υπάρχει στα προϊόντα του PVC. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε και ονομαστική κλίση. 643 μέλη του Κοινοβουλίου συμφώνησαν με την παράγραφο αυτή. Είναι μια, θα έλεγα, πολύ μεγάλη πλειοψηφία και τώρα έχουμε την πρώτη περίπτωση ελέγχου. Μόλιβδο στο PVC και η Επιτροπή λέει εντάξει να κάνουμε περιορισμούς, να επιτρέψουμε όμως κάπως και να επιτρέψουμε ακόμα περισσότερο για τα προϊόντα ανακύκλωσης. Και σύν της άλλης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θέλουμε και μία ετικέτα. Η ετικέτα η οποία θα λέγει ότι ε, πρόκειται για ανακυκλωμένο ε, PVC. Αυτό δηλαδή είναι και θετικό. Ε, γενικά έχεις από τη μία θα έλεγα καινούριο PVC, παρθένο PVC και ανακυκλωμένο. Ο κόσμος θα πει ότι μιλάμε για κυκλική οικονομία και είναι καλύτερο από το καινούριο PVC. Αλλά βέβαια στην ανακυκλούμενη οικονομία το PVC αυτό θα περιλαμβάνει μόλιβδο. Δημιουργούμε και ετικέτες οι οποίες δηλαδή είναι παραπλανητικές. Και συν της άλλης είναι άδικο για όλους αυτούς που έχουν αναπτύξει ήδη εναλλακτικά προϊόντα χωρίς μόλυβδο. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εντελώς λάθος. Έχουμε καταθέσει μαζί με συναδέλφους από Ρινιού και τη σοσιαλιστική ομάδα την αντίρρησή μας μας λέτε ότι υπάρχουν πολλά προϊόντα PVC με μόλιβδο τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι, γι' αυτό θέλουμε να τα ανακυκλώσουμε. Μα ανακυκλώνοντας παρατείνεται το πρόβλημα. Και δεύτερον, και εδώ θα προκαλέσουμε υποτίθεται θέματα στη χημική βιομηχανία. Όταν έρχονται να κάνουν λόμπι, λέγουν ότι στο μέλλον αυτό θα έχουμε χημική ανακύκλωση, ανακύκλωση των χημικών προϊόντων. Εδώ μπορούμε να έχουμε μια λύση, αλλά θα πρέπει να μας δείξουν ότι η λύση αυτή είναι πραγματικά, <clears throat> θα έλεγα, λειτουργική. Η παράταση μέσω της ανακύκλωσης της παρουσίας του μολύβδου είναι κάτι το κακό και γι' αυτό η αντίρρηση που καταθέσαμε έχει νόημα και είναι συμβατή με όλες τις αποφάσεις που έχουμε πάρει μέχρι τώρα σαν Κοινοβούλιο και αυτή της προηγούμενης εβδομάδα. 7 λεπτά. Θα σας δώσουμε λοιπόν το λόγο για 7 λεπτά, καθότι ήσασταν ε, βασικός συντάκτης της αντίρρησης, αλλά παρακαλώ οι υπόλοιποι να μην μακρηγορήσουν τόσο. Η κυρία Ρένα, ευχαριστώ πολύ, πολύ πολύ γρήγορα γιατί τα όσα είπε ο Μπάς είναι πολλά και σημαντικά. Πρώτον, ότι το προαιρετικό μέτρο συχνά αποτυγχάνει. Εμείς θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν πιο δεσμευτικά ε, τέτοια μέτρα ε, και θα πρέπει να ληφθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ανακυκλωμένο PVC, το έχουμε πει εξάλλου. Το γεγονό ότι περιέχουν μόλιβδο αυτά τα προϊόντα με ένα 0,1% συντελεστή ε, δίνει την εικόνα ότι δεν είναι τόσο επιζήμιο, ενώ είναι. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, το να προσανατολίσουμε τον ε, καταναλωτή σε ένα κυκλωμένο PVC μπορεί αυτή τη στιγμή να φαίνεται σαν μια υπεύθυνη ε, στάση και συμπεριφορά σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση του PVC. Όμω ο, ο καταναλωτή αυτό τελικά κατευθύνεται και προσανατολίζεται προ ένα τοξικό προϊόν. Επομένω, πρόκειται για παραπληροφόρηση του καταναλωτή. Και τέλο, το γεγονό ότι υπάρχουν εναλλακτικέ λύσει σε σχέση με αυτέ που προτείνονται σήμερα δείχνει ότι υπάρχουν όλα τα επιχειρήματα προκειμένου να ε, υιοθετηθεί αυτή η αντίρρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μάρτιν Ότσεκ για το Renew. Ευχαριστώ. Τα όσα είπε ο Μπάς, ίσως μόνο σε ένα σημείο θα μπορούσα να δώσω ένα στοιχείο. Αν, αν έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφορετικά, ότι ε, περιέχει ε, επικίνδυνα χημικά. Να επαναλάβουμε όμως ότι δεν υπάρχει ασφαλές όριο για το μόλυβδο. Γιατί και οι επιστήμονε προσπάθησαν να βρουν ένα τέτοιο κατώτατο όριο ασφαλού χρήση και δεν βρήκαν κανένα τέτοιο γιατί έχει να κάνει ιδίω, είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τα παιδιά και την ε, νευρολογική τους ανάπτυξη. Με αυτή την, αντίρρηση, με αυτή την εξαίρεση μάλλον, ε, επεκτείνεται το πρόβλημα και μεγεθύνεται, γιατί πρόκειται για μια απόπειρα ε, να καλύψουμε κάποιο από το Υπάρχουν PVC, να επικαλυφθεί το υπάρχον PVC με δύο άλλες επιστρώσεις ε, άλλου ε, υλικού. Όμως τελικά θα υπάρχει μεγαλύτερη μόλυνση μολύβδου και δεν είναι 0,1, είναι 2% μολύβδου που μπορεί να υπάρχει στο ε, ανακυκλούμενο PVC. Επομένω, πρόκειται εδώ για ένα ζήτημα υπευθυνότητας του παρασκευαστή. Επομένω, ο κλάδο εδώ τη χημία θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε του. Να μην διατηρεί τέτοιου είδου επικίνδυνα υλικά. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα υιοθετήσει αυτή την ε, κυκλική οικονομία, πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν τέτοια παραθυράκια. Γιατί ε, δεν διακινδυνεύεται μόνο η υγεία και το περιβάλλον και μάλιστα εδώ δεν υπήρξε καν μέτρηση των δικτύπων για το περιβάλλον έχει να κάνει με την αποθάρρυνση της κυκλικής οικονομίας. Και εδώ αυτή η εξαίρεση έχει ευρύτερες ε, επιπτώσεις από τη μόνο το περιβάλλον. Και εδώ μιλούμε για 15 έτη, έτσι. Πολύ μεγάλη χρονική περίοδος, απολύτως απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Αλεξάνδρα Μπενχιούμπερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η έκθεση των ανθρώπων στο μόλιβδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μεγάλα βήματα, όμως ε, εμείς εδώ μιλάμε με επιστημονικά στοιχεία. Το ανακτημένο PVC είναι παράγοντας ε, κινδύνου. Χρειάζεται να γίνουν λοιπόν ε, και άλλες αξιολογήσεις, αναλύσεις και μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν γίνει εκτιμήσεις ε, κινδύνου αρκετές για τα διάφορα ε, παράγωγα μολύβδου. Αυτή τη στιγμή το, ο μόλιβδος και τα υποπροϊόντα του είτε καταλήγουν σε κάποια χωματερή είτε καίγονται. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να σκεφτούμε πιο έξυπνους τρόπους διαχείρισης είτε μέσω της ανακύκλωσης είτε μέσω της, της κυκλικής οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν να μετρηθεί η περιεκτικότητα του ανακυκλωμένου PVC σε μόλιβδο μέχρι το 2030 και ε, φυσικά να υπάρχει ανώτατο όριο 0,1% μόλυβδου σε πλαστικό. Αυτό τώρα δεν έχει καμία σχέση με μολύβδινους σωλήνες που είναι 100% από μόλυβδο. Όταν υπάρχει 0,1% ε, μόλιβδο σε έναν πλαστικό σωλήνα, νομίζω πως πρέπει να είμαστε κανεί να δούμε τη διαφορά. Η πρόταση τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι για μας μια αρκετά καλή συμβιβαστική πρόταση, την οποία θα στηρίξουμε. Η πρόταση βέβαια αυτή δεν είναι καλή συμβαστική πρόταση. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Μαντρουά, για τους ECR. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι σε θέση να υποστηρίξω την αντίρρηση. Απορρίπτω το επιχείρημα. μαζί με τα 24 κράτη-μέλη στην Επιτροπή που θεωρούν ότι αυτό το μέτρο είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να δώσουμε το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δοθεί αυτός ο κύκλος ζωής, ανακύκλωση του PVC. Υπάρχουν δύο σημαντικοί αλλά ιδίω παραπληκτικοί ισχυρισμοί. Πρώτον, ότι η επισήμανση προώθησης ε, των ε, υλικών ανακυκλούμενου PVC αντιτίθενται στους σκοπούς ε, του κανονισμού, το οποίο είναι ε, εσφαλμένο, γιατί η επισήμαση παρέχει μια νομοθετική διάκριση μεταξύ ανακυκλούμενου και μη ανακυκλούμενου PVC. Και η Επιτροπή έχει προηγούμενο υπό το πρόγραμμα REACH. Δεύτερον, το ψήφισμα αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ε, και σωστή διάθεση του PVC και ότι, και όλο αυτό ήδη υπάρχει ως υποδομές. Όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να το υποστηρίζουν, υπάρχουν κάποια πιλωτικά προγράμματα, αλλά τίποτα που να είναι εμπορικά βιώσιμο. Επομένως, θα ήθελα να υπενθυμίσω τα συμπεράσματα του Ρίχα Ρέκ, ότι τα όρια και οι εξαιρέσει είναι απαραίτητα γιατί εναλλακτικά θα έπρεπε τέτοιου είδους ε, υλικά ε, ή να πάνε στη χωματερή ή να περάσουν στην καύση στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αντί για την ανακύκλωση, το οποίο θα αύξανε τις εκπομπές, δεν θα μείωνε τους κινδύνους για το περιβάλλον. Αμφιβάλλω ότι θα ήθελαν οι συντάκτε τη αντίρρηση περισσότερη καύση ή περισσότερη χρήση πρώτων υλών. Αυτό ακριβώ θα γίνει όμως, εάν περάσει αυτή η περισσοτερη χρηση πρωτων αυτο ακριβω θα γινει ομως εαν περασει αυτη η αντιρρηση στο Κοινοβούλιο. Υποτίθεται ότι λύνει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, όμως ε, αυξάνει το κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα άλλο και πολύ χειρότερο. Ε, ε, Κλείνοντα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Φλιόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εξωτήμα μέλη. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια τόνοι PVC παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετήσια. Αυξάνονται επίσης και οι εισαγωγέ. Το 10% ε, θα έλεγα ανακυκλώνεται η... Τα νέα προϊόντα βέβαια με PVC ήδη από το 2016 δεν περιλαμβάνουν μόλιβδο. Υπάρχει το θέμα της ρύθμισης του μολύβδου στα προϊόντα εισαγωγής. Υπάρχει το θέμα της έκθεσης των φυσικών προσώπων στο μόλιβδο. Απαγορεύεται επίσης η θέση στην αγορά ε, προϊόντων PVC ε, που περιλαμβάνουν μόλιβδο πάνω από 0,1%. Το ίδιο ισχύει και για τα ανακυκλούμενα προϊόντα PVC στον τομέα των οικοδομών, αλλά οι εξαιρέσεις που υπάρχουν ε, θα πρέπει παρόλα αυτά να προστατεύουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον η ανακύκλωση του PVC είναι ένας πραγματικός τρόπος για μείωση των, της παρουσίας του μολύβδου στο περιβάλλον, διότι καθυστερεί ε, την, ε, θα έλεγα, απόσυψη του προϊόντος. Η χημική ανακύκλωση δεν είναι βέβαια αρκετά ευρεία προς το παρόν για να καλύψει τους στόχους αυτούς. Βρισκόμαστε μόνο σε πιλωτικές φάσεις. Οι εξαιρέσεις στην ουσία που προτείνουμε μας δίνουν κάποιο χρόνο έτσι ώστε να έχουμε καλύτερες τεχνολογίες οι οποίες να είναι πλέον διαθέσιμες. Τα μέτρα που προτείνονται θα μειώσουν το μολύβδο μακροπρόθεσμα στα είδη του PVC και θα περιορίζεται η παρουσία του μολύβδου σταδιακά ώσπου να εξαφανιστεί και να μην χρειάζεται πλέον η ανακύκλωση. Ε, τα μέτρα τα οποία υπάρχουν απαιτούν 675.000 τόνοι PVC που έχουν περισσότερη περιεκτικότητα σε μόλοβδο θα πρέπει να αποσυρθούν. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ε, θα φύγει στο περιβάλλον ένα μεγάλο ποσοστό της μέσω της καύσης ε, του μολύβδου. Είναι, θα έλεγα, ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε να βρεθεί στο περιβάλλον ο μόλυβδος αυτός. Το PVC που περιλαμβάνει LED θα συνεχίσει να εισάγεται χωρίς ε, έλεγχο των επιπέδων ενώ η βιομηχανία έχει σταματήσει να παράγει PVC από το 2016 χωρίς μόλυβδο. Νομίζουμε ότι το μέτρο αυτό και οι εξαιρέσει είναι συμβατές με τους βασικούς στόχους του REACH και βρίσκει μια ισορροπία ανάμεσα στις περιβαλλοντικές ανησυχίες σχετικά με τον παλαιό μόλυβδο και τη χρήση της κυκλικής οικονομίας ε, για το, για PVC. Ακούσαμε τα επιχειρήματα, ακούσαμε και τις παρατηρήσεις σας. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα ε, είναι όμως καλά. Αν ε, θέλετε να καταθέσετε αντίρρηση και είναι δικαιωμά σας, δεν γνωρίζουμε πότε θα υπάρξουν νέα μέτρα τα οποία να υποστηριχθούν από την πλειοψηφία των μελών και από το Κοινοβούλιο. Η πρόταση ψηφίστηκε από 24 μέλη στα πλαίσια της Επιτροπής ΡΙΤΣ. Αυτά ήθελα να πω υπέρ των προτάσεών μας. Θα ψηφίσουμε αύριο για την αντίρρηση. και θα ψηφιστεί την, τον Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Καλώς θα τα πούμε αύριο στις 9. Σε δύο λεπτά ξεκινάει η συνάντηση των συντονιστών. Παρακαλώ μόνο οι συντονιστές στην αίθουσα.